Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να καθίσουμε, να σταματήσουμε τις ατομικές προσωπικές συζητήσεις ο ένας με τον άλλο. Παρακαλώ να διακοπούν οι συζητήσεις μεταξύ ώστε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης δεν έχουμε τροποποιήσεις. Προτείνω να το εγκρίνουμε ως έχει. Στο σημείο 2... Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει web stream το οποίο μας καταγράφει με βίντεο. Έχουμε την κυρία Πετινάρη, την Ιζαμπελ Κλίν. Βρίσκονται στην αίθουσα νέα μέλη. κυρία Πέτινα Νοελιά, Ιζαμπελ Κλίν και Νοηλιά Πετινάρη και χαιρετούμε, αποχαιρετούμε την Κράτια Φιωρέλο. Στο σημείο 3 έχουμε το βασικό σημείο της συνεδρίασής μας. Υποδεχόμαστε ξανά με μεγάλη χαρά τον Επιτροπό μεταξύ μας για μια ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του διαφορετικού διαλόγου. Όπως γνωρίζετε, μιλάμε εδώ για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν για τα έτη 2011-2012 και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 2013. Με λίγα λόγια και με σαφήνεια κύριε Επίτροπε, τι έχει συμβεί, τι κάνουμε τώρα, τι πράτετε τώρα και τι πρόκειται να πράξετε στο μέλλον. Σας δίνω το λόγο για να μας δώσετε μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του τρέχοντος πνεύματος της Κομισιόν ε, όσον αφορά το δικό σας χαρτοφυλάκιο και μετά θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση με τους συναδέλφους. κυρία Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος και το μελλοντικό πρόγραμμα. Στο πρώτο τους πρώτους μήνες αυτού του έτους ε, είδαμε την παράδοση πρωτοβουλειών που εμπίπτουν στο χαρτοφυλλοκιά μου. Ίσως θα μπορούσα να πω και μερικά περισσότερα επειδή από πέρυσι το φθινόπωρο το χαρτοφυλλοκείο των κοινωνικών υποθέσεων της Κομισιόν εστιάστηκε στον κανονισμό για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και μετά μια πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και μετά τη χρήση της πρωτοβουλίας για τις ευκαιρίες και μετά μια πράσινη βίβλο για την αναδιάθρωση της Λευκής Βίβλου για ε, τις συντάξεις και την ε, απόσπαση εργαζομένων και τέλος μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο η δέσμη μέτρων για την απασχόληση επισημάνω και πάλι τα κύρια χαρακτηριστικά των προτάσεων για τις αποσπάσεις που συζητήθηκαν ε, στην περασμένη ώρα ερωτήσεων στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Επίσης αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα, για την υποστήριξη των πολιτικών μετά το 2013, κυρίως το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κομισιόν εγκρίθηκε, εγ, ενέκρινε μια δέσμη μέτρων για την απασχόληση την περασμένη εβδομάδα ε, ενισχύοντας ε, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ήταν απολύτως έγκαιρη αυτή η απόφαση. Μόλις είχαμε λάβει νέα στοιχεία για την επιδείνωση των συνθήκων στην αγορά εργασίας, ε, την αύξηση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη. Στο διάστημα πριν από τη συνεδρίαση αυτή. Θα ήθελα να τονίσω εδώ τρία σημεία στα οποία θα εστιαστεί περισσότερο η Κομισιόν χάρη σε αυτή τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Πρώτον, αυτό το έγγραφο επανακαθορίζει, ευανεστιάζει την προσοχή στην πλευρά ζήτησης της αγοράς εργασίας εστιαζόμαστε συχνά σε πολιτικές που θα δημιουργήσουν ευνοϊκές ε, συνθήκες ε, όπως επιχορηγήσεις ε, πρόσληψης, μεταφορά κονδυλίων και μεταφορά φόρων, υποστήριξη των νεοσυσταθισών επιχειρήσεων και ούτω καθεξής για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και με τη δημογραφική γύρανση του πληθυσμού εστιάζεται η Κομισιόν σε τρεις τομείς. Την πράσινη οικονομία, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και των υπηρεσιών κατοίκων εξυπηρέτησης που παρέχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης. Επίση, ανταποκρίνονται στι κοινωνικέ και οικονομικέ ανάγκε. Προτείνει λεπτομερή σχέδια δράση για την υποστήριξη και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων απασχόληση σε αυτού του τρει τομεί. Σήμερα η αυξανόμενη ανεργία ανησυχεί τους Ευρωπαίους πολίτες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η ανεργία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται. για αυτό το λόγο οι προτάσεις μας για μια δέσμη μέτρων απασχόλησης ε, έρχεται στην κατάλληλη στιγμή καθώς πολλές χώρες υλοποιούν πόδινες μεταρρυθμίσεις ε, πρόσφατα στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Ο πρόεδρο Μπαρόσο παρουσίασε συγκεκριμένε προτάσει για τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ελλάδα. Οι προτάσει μα, ωστόσο αφορούν επίση ε, και μέσω πρόθεσμα ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους στο, πλαίσιο, στο σημερινό πλαίσιο για ευρωπαϊκή δράση ε, με στόχο την επίτευξη των ε, στόχων του 2020. Θέλουμε λοιπόν η αντιμετώπιση της απασχόλησης να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Οι ιδέες που παρουσιάζουμε σήμερα για τα κράτη-μέλη καθώς και οι ενωσιακές δράσεις που παρουσιάζονται καλύπτουν τρεις κυρίους τομείς. Πρώτον, τονίζουμε την ανάγκη να ενισχύσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν βήματα για τη δημιουργία των σωστών συνθήκων, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ζήτησης ε, στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους που ανέφερα προηγουμένως. Ωστόσο, η δέσμη μέτρων εξετάζει επίσης τις διαρθρωτικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη δημογραφική γύρανση, και τις ε, γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αναγνωρίσει τους τρεις τομείς ε, ε, στους οποίους εστιάζονται τα έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο αυτής της δεσμής μέτρων. Πιστεύουμε ότι η επίδραση στην απασχόληση από την επένδυση στις ικανότητες σε αυτό το τομέα είναι σημαντική. Ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθούν 20 εκατομμύρια θέσει εργασία μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την υποστήριξη και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων απασχόληση σε αυτού του τρει τομεί. Δεύτερον, πρέπει η αγορά εργασία στην Ευρώπη να γίνει πιο δυναμική. Βάσει των διδαγμάτων που έχουν αποκομιστεί από την πλέον παρατεταμένη κρίση, η Κομισιόν προτείνει στα κράτη-μέλη να επενδύσουν στην επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασία. Για τη δημιουργία θέσεων εργασία πρέπει οι αγορέ εργασία να γίνουν πιο δυναμικέ και χωρί αποκλεισμού. Αυτή η ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί μέσω πολιτικών απασχόληση που καθιστούν πιο ευέλικτε τι χώρε εσωτερικά με μείωση του φορολογικού κόστου και τη αβεβαιότητα με την υποστήριξη των βιώσιμων συνθήκων και την αποφυγή των παγίδων για την καταπολέμηση της κατάτμισης της αγοράς εργασίας. Η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει την ποιότητα των εργασιών με μια δημόσια διαβούλευση για ένα ποιοτικό πλαίσιο για, τις, ε, ε, για τα προγράμματα εκπαίδευσης. Συγκέντρωση των πόρων και αποτελεσματικές εταιρικέ σχέσεις είναι απαραίτητες για τη σωστή υλοποίηση οποιασδήποτε πολιτικής απασχόλησης. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας πρέπει να λαμβάνουν χώρα παράλληλα με επενδύσεις σε ανθρώπους. Η επένδυση λοιπόν σε ικανότητες είναι επίσης κρίσιμη σημασία για την αντιμετώπιση της έλλειψης ε, δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας ε, γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης ε, της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων και αποφυγής της ασυμφωνίας μεταξύ ε, δεξιοτήτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, για να βελτιωθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη πρέπει να άρουμε τα οποιαδήποτε νόμιμα και πρακτικά εμπόδια που υπάρχουν όπως, ε, με διάφορα μέτρα όπως η φορητότητα των συντάξεων για παράδειγμα. Επίσης προτείνουμε να αλλάξουμε το σημερινό εργαλείο Γιούρε, ώστε να ε, βρίσκει τις συμφωνίες μεταξύ δεξιοτήτων, μεταξύ των κρατών μελών τρίτων, το ιδέσμι μέτρων για την απασχόληση, προτείνει τρόπους ενίσχυσης του συντονισμού και της πολυμερούς παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου το πίνακα αποτελεσμάτων scoreboard για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όσον αφορά την ανεργία. Οι εταίροι θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο στον ορισμό προτεραιοτήτων και στη χάραξη πολιτικών. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε τη συμμετοχή των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την παρακολούθηση των εξελίξεων. Πρόταση είναι ενίσχυση της διακυβέρνησης σε ενωσιακό επίπεδο, ενισχύοντας και τις επιτόπου ε, διακυβερνήσεις. Οι δέσμοι μέτρων για την απασχόληση θα τεθεί σε ισχύ το επόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Επίσης, το πακέτο αυτό ενισχύει και τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ των μεταρρυθμίσεων, των ε, επενδύσεων για την υποστήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά θέλω να σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα το πρόγραμμά μας για το υπόλοιπο του 2011 που ήδη έχουμε παρουσιάσει στον νομοθέτη και που αφορά κυρίως ε, τα μέτρα για την απόσπαση εργαζομένων. Στην ώρα ε, ερωτήσεων της περασμένης εβδομάδας ακούσαμε πολλές ερωτήσεις από πολλούς συναδέλφους σε σχέση με τις προτάσεις της Κομισιόν της 21ης Μαρτίου. Ο σκοπός αυτής της συνεδρίασης δεν είναι να επαναλάβουμε τι ιδιε ερωταπαντήσεις, ερώτα-απαντήσει, να έχουμε την ίδια συζήτηση σε σχέση με το περιεχόμενο των προτάσεων. Απλά ήθελα να υπενθυμίσω τα τρία κύρια χαρακτηριστικά. Με αυτέ τι προτάσει, η Κομισιόν εκπληρώνει μια υπόσχεση του έγινε από τον πρόεδρο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009 να επιλύσει τα προβλήματα που αφορούν την ερμηνεία και την υλοποίηση της οδηγίας απόσπασης εργαζομένων. Έτσι επιτυγχάνονται ισορροπίες σε πολλά επίπεδα τηρούνται οι στόχοι της οδηγίας του 1996, τηρούνται οι διαφορετικοί χαρακτήρες των διαφορετικών κοινωνικών μοντέλων, αποφύγει ε, περί του διοικητικού φόρτου το πακέτο, περιλαμβάνει μια οδηγία εκτελεστική για την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας του 1996 για την απόσπαση των εργαζομένων και επίσης ένα κανονισμό για τη διευκρίνηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών μαζί με τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Η πρόταση για ένα κανονισμό επιβεβαιώνει ότι δεν θέλουμε να εμποδίζεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης ε, ε, σε σχέση με το δικαίωμα απεργίας και αντίστροφα δεν θέτει επιπλέον φραγμούς για το δικαίωμα απεργίας. Η εκτελεστική οδηγία θέτει πιο φιλόδοξα πρότυπα για την απόσπαση εργαζομένων και για τις εταιρείε όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Καθιερώνει κανόνες συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών όσον αφορά τις αποσπάσεις, διευκρινίζει τις, ε, τα στοιχεία της έννοιας της απόσπασης ώστε να αποφεύγεται η ο πολλαπλασιασμός εταιριών που χρησιμοποιούν την απόσπαση για να παρακάμπτουν τον νόμο καθορίζει ευθύνες όσον αφορά τις επιθεωρήσεις και διευκρινίζει τα μέτρα εθνικού ελέγχου, βελτιώνει την ενίσχυση της εφαρμογής των δικαιωμάτων με έναν μηχανισμό ε, υπευθυνότητας και ε, βοηθάει την επιβολή διασυνοριακών προστήμων και κυρώσεων. Κάθε αρχείο αφορά μια πρόταση και το προτινόμενο πακέτο είναι το πιο αποτελεσματικό για την προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων και το πιο αποτελεσματικό ως προς το κόστος, τόσο για τις εταιρείε όσο και για τα κράτη. Οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στο άτυπο Συμβουλίο μεταξύ Υπουργών Απασχόλησης Αναμένω με αγωνία την πρόταση και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και για τις δύο αυτές πρωτοβουλίες. Τώρα θα περάσω στο χρηματοπιστωτικά μέσα, στα δημοσιονομικά μέσα. Όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις για τις προτάσεις της Κομισιόν βρίσκονται υπό εξέλιξη. Γνωρίζω ότι ξεκινήσατε να μελετάτε διάφορες προτάσεις και ότι πολλά σημεία ήδη συζητώνται ένθερμα. Ε, η παράκληση που θα ήθελα να κάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι να μην ξεχνάμε την κρίσιμη σπουδαιότητα της είδηση των δημοσιονομικών μας μέσων με τους πολιτικούς μας στόχους και την ικανότητά μας να δημιουργούμε πραγματική προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν έχει προτείνει ένα ελάχιστο μερίδιο που να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 84 δισεκατομμύρια ευρώ του κονδυλίου για το Ταμείο Συνοχής να δοθούν στο Κοινωνικό Ταμείο. Στο Συμβούλιο πολλά κράτη-μέλη έχουν δείξει την υποστήριξή τους για αυτή την πρόταση, ωστόσο άλλα κράτη αντιτέθηκαν στεναρά. Καταλαβαίνω τις ε, διαφορετικές αποφάσεις ε, και που ακούστηκαν και στο Κοινοβούλιο για αυτό το σημείο. Θα ήθελα να επανέλθω εν συντομία στην λογική που υποστηρίζει αυτή την πρόταση. Το να έχουμε ένα προκαθορισμένο μερίδιο του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υποστηρίζουμε την κοινωνική χωρίς αποκλεισμούς ε, πτυχή της ανάπτυξης αποτελεί μια αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει σοβαρά τα όσα υπόσχεται και ότι αφιερώνει κάποιο κομμάτι του προπολογισμού σε αυτά δεδομένη της τρέχουσας κατάστασης επιβάλλεται να συγκεντρώσουμε τους οικονομικούς μας πόρους ώστε να ε, βάλουμε ανθρώπους να εργαστούν, να βρούμε δουλειά σε ανθρώπους. Το κυριότερο πρόβλημα εδώ είναι η αυστηρότητα. Θα μειωνόταν η ευελιξία των κρατών μελών να αποφασίζουν πόσα θα ξοδεύουν στα κοινωνικά προγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το επιχείρημα δεν είναι έγκυρο. Τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για όλα τα δημοσιονομικά μέσα, όπως το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, ε, πρέπει να έχουν ελάχιστα ποσά τα οποία αιτιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Αρχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι θα υλοποιηθούν. Αν δεν αναστρέψουμε την καθοδική πορεία που έχουμε σήμερα, ο στόχος της κοινωνικής Ευρώπης δεν θα μπορέσει να είναι αξιόπιστος. Τα ελάχιστα μερίδια που προτείνουμε βοηθούν τα κράτη-μέλη να έχουν την ευελιξία να προσαρμόσουν τα κονδυλιά τους στις επιμέρους ανάγκες τους. Ε, τα ελάχιστα μερίδια που προτείνουμε δεν είναι αδύνατα, ανέφικτα για τα κράτη-μέλη στις περισσότερες περιπτώσεις. Ε, είναι πολύ κοντινά στην τρέχουσα κατάσταση και θα έχουν από αποτέλεσμα ελάχιστη αύξηση σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Σε ορισμένα κράτη-μέλη ωστόσο η κατανομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Συνοχής κοινωνικού ταμείου αποτελεί 10-15% αύξηση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο από αυτά θα ε, ε, επενδυθεί σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τουλάχιστον κατά ένα ελάχιστο ποσοστό. Το να ορίζουμε τα ελάχιστα μερίδια σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο παρέχει απόλυτη ελευθερία στις εθνικές αρχές, ανεξαρτήτως των στόχων του 2020, να επιλέγουν πόσα κονδυλία θέλουν να επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Είμαι πεπισμένος ότι η Επιτροπή σας συμφωνεί με τον πολιτικό στόχο της Κομισιόν και υπολογίζω σε εσάς να δώσετε την υποστήριξή σας για αυτό το συγκεκριμένο μέρος της πρότασής μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το Κοινοβούλιο να διασφαλίσει κατά την νομοθετική διαδικασία ότι θα διατηρηθούν τα ελάχιστα μερίδια ώστε πραγματικά να μπορούμε να μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό για την κοινωνική Ευρώπη. Αυτό φυσικά λειτουργεί παράλληλα με όλα τα στοιχεία των προτάσεών μας που έχουν στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τώρα να πω λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Δεν θα πρέπει, πιστεύω, να πείσω την Επιτροπή σα για την προστιθέμενη αξία αυτού του εργαλείου. Είναι απαραίτητο για να καταδείξουμε την ελληνική που έχουμε έναντι αυτών που αντιμετωπίζουν σοβαρέ δυσχέρειε. Είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να δοκιμάσουν καινοτόμε προσεγγίσεις και να βοηθήσουν ανθρώπου που προσπαθούν να βρουν εργασία. Είναι ένα τρόπο για να δείξουμε ότι η Ευρώπη έχει νόημα. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε δυσκολίε στα επιμέρου σημεία τη πρόταση και είμαι ανοιχτό να συζητήσουμε περαιτέρω δυνατέ βελτιώσει. Όμω, σα παρακαλώ να μα στηρίξετε και να υποστηρίξετε αυτό το εργαλείο το οποίο θα κάνει μια μεγάλη διαφορά και για τους μονομένους ανθρώπους, αλλά για το πώς βλέπουμε γενικότερα την Ευρώπη. Κατανοώ ότι το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Είναι να εξελίξει τήσεις στο Συμβούλιο και μπορεί σύντομα να υπάρξει και συμφωνία. Στα πλαίσια του Συμβούλου δεν θα μπω σε λεπτομέρειες προκειμένου, καθώς εσείς ακόμη δεν έχετε ε, ολοκληρώσει την θέση σας. Απλά να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το εργαλείο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκκινήσει δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, επίσης, υπάρχουν κάποιες προτάσεις για την κατανομή κονδυλίων μέσα από αυτό το εργαλείο και αυτό θα γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι κάτι λοιπόν που θα πρέπει να μιλήσουμε πολύ προσεκτικά ε, και να πω τέλος ε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ότι η συζήτηση για το πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013 ήδη έχει ξεκινήσει και είμαι εδώ όλο αυτιά για να ακούσω τι προτάσει σα. Η αλήθεια είναι ότι το 2013 θα είναι μια χρονιά με όχι λιγότερες προκλήσεις από το 2012 υπάρχει το δυναμικό μέσω των προτάσεων που ήδη έχουμε υποβάλει να αλλάξουμε ε, σημαντικά το τοπίο. Επίσης είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στο έτοιμά σα για την υποβολή μιας πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης ε, του όλου οικοδομήτους μέσω επενδύσεων ταυτόχρονα. Υπάρχουν και πολλές άλλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που φορούν τους Ρωμά, την φορητότητα των συνταξιδικών δικαιωμάτων, την ενεργό συμμετοχή, δημογραφικά στοιχεία, διγύρνους του πληθυσμού, λέω μεταξύ άλλων. Αλλά και πάλι καλύτερα θα ήταν να σταματήσω εδώ και να ακούσω τις δικές σας ε, προτάσεις και να κάνω ό,τι μπορώ για να σας απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Με την παρουσίασή σας μας δίνετε ήδη μία εικόνα του πόσο πυκνές είναι οι προτάσεις που έχουμε μπροστά μας αλλά και του εύρους του χαρτοφυλακίου σας και της αλληλεπίδρασής του με άλλες δράσεις και άλλες πολιτικές που υλοποιούν και μελετούν άλλα μέλη της Επιτροπής. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε εμείς το διαφρομένο διάλογο και θα ήθελα να δώσω πρώτα απ' όλα το λόγο στο συντονίστη κύριο Τσαμπαόρη για την ομάδα ΕΛΚΑ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές φορές ε, έχουμε εκφράσει τη δυσαρέσκειά μας όσον αφορά το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λέγοντας ότι οι βουλευτές θέλουν να δουλέψουν και οι προτάσεις δεν έρχονται, δεν φτάνουν μέχρι εμάς. Ε, εδώ λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον κύριο Επιτροπό που βρίσκεται εδώ. Είναι πολύ χρήσιμο η παρουσία του εδώ και έτσι οι προτάσεις έρχονται και σε εμά και έτσι μπορούμε τόσο να τις επικρίνουμε αλλά και να ευχαριστήσουμε που μας τις παρέχεται κάποιες ερωτήσεις, έχω κάποιες ερωτήσεις για εσάς, χωρίς να θέλω να ε, πάρω όλο το χρόνο και να εμποδίζω τους υπόλοιπους βουλευτές από το να μιλήσουν. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε αυτή τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, τις διάφορες προτάσεις. Ε, έχουμε διάφορες ιδέες, το ίδιο έχετε και εσείς, ε, ιδέες για προτάσεις. Θα τις συζητήσουμε. Μας ανησυχεί λίγο το γεγονός ότι αυτές οι προτάσεις θα πάνε στο Συμβούλιο λίγο νωρίς. Ωστόσο θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια θέση, μια άποψη. Δεν ε, μας είναι απολύτως ε, σαφές πώς θα γίνει η υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Πρόκειται για εθνικές εξουσίες, ε, να ελπίζουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα δημοσιονομικά ζητήματα. Ακούγοντάς σας κύριε Επίτροπε, καταλαβαίνετε καλά τα προβλήματά μας. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες. Αν όμως δεν υπάρχουν χρήματα, αν δεν υπάρχουν κονδύλια, τότε ε, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα πρέπει να βρουν τα κονδύλια ε, βάσει των προτεραιοτήτων τους. Ε, δηλαδή το όλο πράγμα θα υλοποιηθεί βάσει των δημοσιονομικών δυνατοτήτων των κρατών μέλων. Σε ορισμένες χώρες η κατάσταση είναι καλύτερη, το ίδιο και η απασχόληση βρίσκεται σε καλύτερα επίπεδα. Σε άλλες όμως χώρες δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για την ένταξη και υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Η σύνδεση με την πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική, το έχουμε συζητήσει ήδη. Όταν μιλούσαμε για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, εκείνη την εποχή μας είχατε πει ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε το πόσο σπουδαία είναι η πολιτική απασχόληση. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμόντα ερωτήματα. Όσον αφορά την απόσπαση των εργαζομένων, συμφωνώ επί της αρχής. Έχω την εντύπωση ότι οι κανόνες είναι υπερβολικά πολλοί. Υπερβολικά πολλοί έλεγχοι, υπερβολικά μεγάλη γραφειοκρατία. Αυτές οι προτάσεις ωστόσο έχουν έρθει πλέον στο Κοινοβούλιο και θα τις συζητήσουμε ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά το τη δύο θα πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει εμείς να πούμε τις απόψεις μας, τόσο το Συμβούλιο θα λάβει τις αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιτευχθεί συνένεση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σημεία, η κυρία Ελίζαμπετ Μωρά ε, θα μιλήσει για το Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Θα μιλήσει η κυρία Μπάουερ. Ναι, ε, κύριος ε, Αλέξανδρος Σιρκας και, με... και μετά η κυρία... Κύριο Σέρκας, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Αν δεν κάνω λάθος στοιχεία μου, είναι η τρίτη φορά που έχουμε τη χαρά να σας έχουμε μαζί μας Πρώτα απ' όλα στην Ολομέλεια, έπειτα στη συνεδρίωση των ιστών και σήμερα στην Επιτροπή μας. Ελπίζω αυτό να είναι ένα δείγμα της αλλαγής που δείχνουμε στη στάση από πλευρά των Επιτρόπων να μας παρουσιάζουν το σύνολο των εργαλείων της κοινωνικής πολιτικής και τον θεσμικό ρόλο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κοινοτικό μοντέλο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την διαθεσιμότητά σας να μας ακούτε προσεκτικά. Κύριε Επίτροπε και σας παρακαλώ να διαβιβάστε και στους αδέλφους σας ότι πέρα από το να μας ακούτε να μας προσέχετε και λίγο περισσότερο, γιατί καλό να μας ακούτε, αλλά να μας προσέχετε λίγο περισσότερο είναι σημαντικό. Μιλώ εξ ονόματος ε, της ολιστικής ομάδας και πιστεύω ότι πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές που μπορεί να έχουμε, πέρα από τις διαφορές που μπορεί να έχουμε στο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα, τη σήμερα ημέρα, υπάρχει απόλυτη ομοφωνία ότι ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει δεν οδηγεί πουθενά, παρά μόνο σε πιο πολλά κοινωνικά προβλήματα, περισσότερη ανεργία και περισσότερο κοινωνικό αποκλεισμό. Κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι έχει φτάσει η στιγμή να έχουμε μια πραγματική αλλαγή. Όχι αλλαγή μόνο στη φιλοσοφία που βλέπουμε στο πακέτο για την απασχόληση, αλλά μια ουσιαστική αλλαγή, πρακτική αλλαγή για τα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση, την ποιότητα στην απασχόληση, για την ανάπτυξη. Φοβούμαι ότι όλα αυτά ήδη τα έχετε εκφράσει, αλλά μόνο θεωρητικά. Όλα είναι λόγια ακόμη. Δεν βλέπω δηλαδή πρακτικά πώς αυτά τα λόγια θα γίνουν πράξη. Δεν υπάρχει αν θέλετε ακόμη νομοθετική ε, πρόταση ε, τέτοια που να γίνει και εκτιμένο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, την ανεργία που έχει σε τραγικά διέξοδα σε κάποια κράτη-μέλη. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας υποστηρίζουμε για την όλη αλλαγή στη στάση σας, την πολιτική και ιδεολογική αλλαγή που δείχνετε ως μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει πρακτικά να κάνουμε πράγματα για να βελτιώσουμε την κατάσταση ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κύριε Επίτροπε, όλα αυτά που λέμε είναι ενδιαφέροντα, αλλά τι νόημα έχουν στα αυτιά ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 20% ανεργία γενικά και 40% ανεργία μεταξύ των νέων. Είπατε ότι θα υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη. Και το πρώτο που έχω να σας πω είναι το εξή. Θα πρέπει να υπάρχει ακολουθία ανάμεσα στην κοινωνική πολιτική που υποστηρίζει τους κοινωνικούς στόχους και την οικονομική και φορολογική πολιτική. Διότι ενώ από τη μία πλευρά λέτε θα υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη και καλείται τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν συμβουλές για τις δημοσιονομικές δαπάνες. Από την άλλη έχουμε μια φορολογική και δημοσιονομική πολιτική που τρέχει μόνο πίσω από το δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν μπορεί σίγουρα να επιτυχεί αυτούς τους κοινωνικούς στόχους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στην δημοσιονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Ιδάλλως δεν θα κάνουμε τίποτα. Η Ευρώπη ιδάλλως δεν μπορεί να βοηθήσει. Να κλείσω κύριε Επίτροπε γιατί υπάρχουν και άλλοι σοσιαλιστές συνάδελφοι που θα το λόγο. Το κοινωνικό πακέτο που μας παρουσιάσετε σήμερα είναι πολύ καλό αρκεί να υπάρχει ακολουθία με την οικονομική διακυβέρνηση, χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις και ανακολουθίες ανάμεσα στα λόγια και στι πράξει. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ακολουθία ανάμεσα στι θέσει όλων. Και κλείνοντα. γιατί άλλοι συνάδελφοι θα μιλήσουν για την κινητικότητα των εργαζομένων, θα κλείσω με κάτι πιο ε, φιλικό απέναντί σας. Η ομάδα μας θα σας υποστηρίξει απόλυτα σε ό,τι αφορά το Ταμείο για την ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, θέλω να πω ότι αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Σε μια εποχή ε, τεράστια κρίση στην Ευρώπη, το μόνο ήπιο εργαλείο που υποστηρίζει που στηρίζουν τους, κρίσεις, ε, τους τομείς ε, σε κρίση, είναι πολύ σημαντικό. Ε, ας μην το απαξιώνουμε, χρησιμοποιώντας το για άλλους λόγους, παρά για αυτούς που είναι οι βασικοί για να μπορέσουν οι ε, εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα να βρουν μια νέα θέση εργασία. Η κυρία μετά θα Κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο θέματα. Πρώτο, το ESF, ο Μηχανισμό Σταθεροποίησης. Δύσκολο μου φαίνεται αυτό το 25% ως στόχος για να αγωνιστούμε. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες συμμαχίες, κυρίως μεταξύ των Υπουργών Απασχόλησης, που ε, είναι και αυτοί οι οποίοι θα προωθήσουν τα έργα. Αλλά αν αφήσουμε τον κανονισμό του ESF όπως είναι, δεν θα μπορέσει να γίνει. Διότι ο κανονισμός προβλέπει στο άρθρο 4 μια συγκέντρωση που σημαίνει ότι στην ουσία δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί. Κάτι δηλαδή το οποίο να σημάνει σωστή κοινωνική πολιτική απασχόλησης και συμπερίληψης. Και γι' αυτό σα παρακαλέσω κύριε Επίτροπε να δείξετε, να επιτρέψετε να υπάρξει περισσότερη ευκαμψία. Τότε θα βρεθούν και οι συμμαχίε. Το δεύτερο, για την Enforcement Directive, για σχετικά δηλαδή με την ε, οδηγία απόσπαση εργαζομένων. Λέτε εκεί ότι σε ό,τι αφορά τα εθνικά μέτρα επιθεωρήσεων, ότι θέλετε να ξεκαθαρίστε το τοπίο. Όμω στην πραγματικότητα θέλετε να τα περιορίσετε. Είπα εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα τι σημαίνει έστω και ο μικρότερο περιορισμό. Αμέσω το κενό που θα δημιουργηθεί θα προσπαθήσουν να το καλύψουν διάφοροι εγκληματίε και να ε, μειώσουν του μισθού των εργαζόμενων. Γιατί θέλετε να περιορίσετε τι εθνικέ επιθεωρήσει, πιστεύετε πραγματικά ότι με ένα σύστημα IEM είναι δυνατόν αυτό να υποκατασταθεί στους εθνικούς επιτόπου ελέγχους οι οποίοι πραγματικά πρέπει να είναι πολύ αυστηροί. Thank you much. Σας ευχαριστώ. Για την δέσμη μέτρων για την απασχόληση. Χαίρομαι που και εσείς το βρίσκετε επίκαιρο, επίκαιρη τη δέσμη δηλαδή και συμφωνώ με τον κύριο Σέρκας για την ανάγκη συμφιλίωσης των κοινωνικών πολιτικών και της απασχόλησης και των οικονομικών πολιτικών από την άλλη. Αυτή η συμφιλίωση δεν μπορεί να γίνει βέβαια μέσα στην ίδια τη δέσμη μέτρων. Θα πρέπει να γίνει μετά από την έγκριση της δέσμης και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι η δέσμη αυτή θα περάσει και στο εργασίο και του, συνεργασία μάλλον και του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα συμπεράσματά του της 1ης Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε το ίδιο πράγμα και ελπίζω ότι το Συμβούλιο Υπουργών δηλαδή και ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό της ε, ατζέντα και ελπίζω η δέσμευτη να μπορέσει να αποτελέσει την βάση για μια διαφορετική πολιτική και μια διαφορετική στρατηγική που να είναι ένας πραγματικός βιώσιμος τρόπος για να ξεφύγουμε από την κρίση. Όλα τα στοιχεία κλειδιά περιέχονται σε αυτήν. Ανταποκριθήκαμε στις αδυναμίες και ελλείψεις της ε, στρατηγικής για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν ε, κυρίως ε, βασισμένη σε μέτρα για την πλευρά της προσφοράς Έχουμε λάβει υπόψη και τα άλλα δεδομένα της ε, απασχόλησης. Προσφέρουμε δε περισσότερα μέσα, περισσότερα εργαλεία υπέρ της κινητικότητας για να στηρίξουμε τους νέους ε, κυρίως εργαζόμενους που αναζητούν απασχόληση σε άλλη χώρα Θα χρειαστεί λοιπόν να δουλέψουμε πάνω στη δέσμη αυτή, όχι μόνο για την εφαρμογή στον τομέα της απασχόλησης, αλλά και με τρόπο ευρύτερο για τις γενικότερες, ευρύτερες οικονομικές πολιτικές. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Θα χρειαστεί βέβαια να υπάρξουν και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις και ανακατανομές στην τρέχουσα περίοδο και αυτά τα στοιχεία ήδη έχουν αντιμετωπιστεί στην πρωτοβουλία ίσων ευκαιριών που μπαίνει στην φάση της εφαρμογής της. Έχουμε μιλήσει ήδη και έχουμε βάλει τα σχετικά θέματα και μέσα στο πακέτο της απασχόλησης, αλλά θα δώσουμε και περαιτέρω πληροφορίες, καθώς τα, οι ομάδες δράσης θα επιστρέφουν στις 8 χώρες όπου γίνονται οι ανακατανομές για την απασχόληση ιδίως των νέων. Αυτό βέβαια δεν είναι συμπτωματικό, το γεγονό ότι τονίζουμε τη σημασία των δημοσιονομικών εργαλείων για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική. Σημείωσε και το όσα η κυρία Σουρέντερ για την ανάγκη ευκαμψίας. Και όταν το MFF φτάνει στην περίοδο της εφαρμογής θα χρειαστεί κάποια ευκαμψία, δηλαδή το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά σε αυτό θα χρειαστεί να τονίσουμε και περισσότερα επιχειρήματα και να εξοπλίσουμε καλύτερα την αρχική πρόταση που κάναμε για να δώσουμε και την πλήρη αιτιολόγηση των μέτρων και των λύσεων που προτείνουμε και αργότερα θα δούμε που μπορεί να είναι θεμητό να μπουν στοιχεία ευκαμψίας χωρίς να υπονομευθούν οι στόχοι. Σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων για, τη, για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, όπως είπε ο κ. Σωρή, ελπίζω ότι καταφέραμε να μειώσουμε, να περιορίσουμε τα, τις απαιτήσει στις απολύτως απαραίτητες, στο απολύτως απαραίτητο επίπεδο. Και γι' αυτό πήραμε μόνο ένα κλάδο της οικοδομής, όπου βρήκαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα και όπου είναι απαραίτητο να αναλυφθεί νέα δράση και να προταθούν νέες λύσεις, αν θέλουμε να εξαλείψουμε τις προβληματικές περιοχές και τις αμφιλεγόμενες πτυχές, κατά τα άλλα, δεν επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά, με περιττρό τρόπο δηλαδή την αρχική οδηγία. Τώρα βέβαια είναι περιορισμένη η έλεγχη, επιθεωρήσεις. Το είπα ήδη αυτό στην, Ευρωπή, στην Ευρωβουλή μετά από την ερώτηση της κυρίας Τούρουνεν για το ίδιο θέμα ότι οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για να συμμορφωθούμε απόλυτα με το κοινοτικό δίκαιο. Δεν έπαιξε ρόλο απολύτως καμία άλλη σκέψη ή προβληματισμός. Ευχαριστώ. Για το δεύτερο γύρο τώρα. Η κυρία Μωρά Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ ξανά ενώπιον της Επιτροπής μας για να παρουσιάσετε τη δέσμη μέτρων σας και για να τη συζητήσετε μαζί μας. Όπως είπε ένας συνάδελφος πριν από μένα, τόσο όσο ενδιαφέρουσα είναι η φιλοσοφία, τόσο χρειαζόμαστε σήμερα πρακτικές προτάσεις. Χρειαζόμαστε αυτή η δέσμη μέτρων για την απασχόληση να φέρει αποτελέσματα και να αλλάξει την κατάσταση η οποία είναι δυσβάσταχτη σήμερα με την αύξηση της ενεργείας ε, σήμερα στις ευρωπαϊκές χώρες. για αυτό το λόγο θα σας κάνω τέσσερις ερωτήσεις και θα σας κάνω και μια πρόταση. Η πρώτη ερώτηση αφορά τη ζήτηση. Μιλήσατε για ζήτηση μέσα σε αυτό τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση στην οποία βασίζεστε. Ζήτηση στην αγορά εργασίας. Σήμερα πιστεύω πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε αποτελεσματικοί σε κάθε κλάδο, σε κάθε επαγγελματικό κλάδο θα πρέπει να λάβει χώρα ένας πραγματικός προβληματισμός θα πρέπει να καθορίσουμε τις προδιαγραφές, τις αναμένες προδιαγραφές για τις θέσεις απασχόλησης. Επειδή αυτό που βλέπουμε πραγματικά στην αγορά είναι ότι στους επαγγελματικούς τομείς δεν γνωρίζουμε καλά που οδεύουμε. Πρέπει να περιγράψουμε σωστά τις προδιαγραφές των θέσεων που ζητούνται ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε κατάρτιση, επαλήθευση των εμπειριών και των ικανοτήτων, ώστε να καλύψουμε την ζήτηση. Το δεύτερο σημείο μιλήσατε για τρει στόχου πράσινη οικονομία, τεχνολογίες ε, επικοινωνιών και πληροφορικής και υπηρεσίες. Το βλέπουμε καλά στο ότι υπάρχει εξέλιξη των ε, θέσεων εργασία. Και αυτέ αφορούν όλου του κλάδου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί διαφορετικά θα έχουμε επαγγελματικού αποκλεισμού. Το τρίτο σημείο, το υπογραμμίσατε, είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για του νέου. Είπατε ότι θέλετε η πολιτική σας να αντιμετωπίσει αυτό το ευαίσθητο σημείο και ο κ. Σέρκας είπε, ε, ανέφερε πόσο η ανεργία πλήττει τους νέους σήμερα δεν θα το λύσουμε αναπτύσσοντας απλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν την ένταξη στον επαγγελματικό κόσμο. Συχνά χρησιμοποιήθηκαν νέοι για εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς αύριο. Τέταρτο σημείο για το οποίο ήθελα να μιλήσω είναι η, η των κεκτημένων δεξιοτήτων. Θα ήθελα να σας προτείνω κύριε Επίτροπε παρατηρούμε στην εθελοντική εργασία, στις εθελοντικές ενώσεις, να αναπτύσσονται πολλές δεξιότητες. Καμία από αυτές δεν επικυρώνεται στον τομέα του εθελοντισμού. Επικύρωση η οποία θα επέτρεπε μια κινητικότητα για την οποία μιλήσατε, μια εξέλιξη στη διαδρομία. Ας ανοίξουμε λοιπόν αυτό το φάκελο και ας επιτρέψουμε να υπάρχει τέτοια επικύρωση η οποία θα επιτρέψει την εξέλιξη των ανθρώπων που έχουν εργαστεί στον εθελοντισμό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στίβεν Χιούζ και μετά ο κύριος Πάγος. Στίβεν Χιούζ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τη μάχη που συνεχίζεται να δίνεται για την κοινωνική πολιτική, ιδίω θεσμικά όργανα που είναι πολύ εχθρικά προ την κοινωνική πολιτική κάνω δύο σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα για το πακέτο για την απασχόληση. Συμφωνώ με τα σχόλια που ήδη ακούστηκαν και δεν διαφωνώ με την ανάλυση που κάνει σε αυτό το πακέτο και χαιρετίζουμε αυτό το πακέτο σε σχέση με τη γλώσσα που ακούγεται σχετικά με την εξέλιξη τη μακροοικονομική διακυβέρνηση όπω ακούγεται τελευταίου μήνε. Αυτό όμω που δύσκολα κανεί ε, ε, μπορεί να παραγνωρίσει είναι ότι δεν διαφέρει σημαντικά αυτή η ανάλυση με τι κατευθύνσει γραμμέ στην απασχόληση του 1997. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η στρατηγική του 1997 είχε οδηγήσει σε συγκεκριμένες οδηγίες για τη μερική απασχόληση ε, και για ε, την ε, απασχόληση των συμβασιούχων. Και είναι μια σημερινή στρατηγική που οδήγησε σε άτυπες μορφές απασχόλησης και κατανοήσαμε ότι ήταν μια επικίνδυνη τάση γιατί αυτό οδηγούσε σε μείωση των προτύπων εργασία, και άρα λοιπόν τα δείγματα είναι ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη βάση, ε, ένα σταθερό πυρήνα προτύπων για την απασχόληση και χρειάζεται λοιπόν μια οδηγία σε κοινωνικό επίπεδο που να θεσπίζει αυτά τα πρότυπα. Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό, δηλαδή με βάση την αλήθεια που έγινε το 1997 και τα διδάγματα που αντιλήσαμε τότε. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό σήμερα, για ποιο λόγο. Δεύτερο σχόλιο για το πακέτο απόσπαση εργαζομένων. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια, αλλά είπατε και σήμερα κάτι που αναφέρατε και στην Ολομέλεια, ότι η πρότασή σας δεν θεωρεί ότι προέχει το δικαίωμα για την παροχή υπηρεσιών, ούτε ε, επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα ε, του συνεταιρίτες και ότι προσπαθεί να ξέρετε μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων. Ε, το δικαίωμα στην απεργία και το δικαίωμα στον συνδικαλισμού είναι δικαιώματα στο, στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ούτως ή άλλω. Το δικαίωμα της εγκατάστασης αντίθετα και το δικαίωμα της επιχειρήσεων δεν είναι δικαιώματα που περιέχονται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε πώς μπορούμε να μιλάμε για απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στα δύο. δηλαδή τα δικαιώματα που αφορούν τις επιχειρήσεις, δεν είναι κομμάτια του α, πρωτογενούς δικαίου, όπως τα δικαιώματα στο συνδικαλισμό και στην απεργία. Και ρωτώ λοιπόν γιατί κάνετε αυτή την εξίσωση στην πρότασή σας. Ε, Edith Bauer και στη συνέχεια για το Εκτός ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να σημειώσω με ενδιαφέρον την αλλαγή παραδείγματος, διότι μέχρι τώρα είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε επενδύσει για την απασχόληση, για να ικανοποιήσουμε την ζήτηση. Διαπιστώνω τώρα μια εξέλιξη στην, ε, στον τρόπο αυτό σκέπτεστε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα τώρα και από τη σκοπιά της ζήτησης. Νομίζω ωστόσο ότι αυτό μπορεί να σημαίνει νέες προκλήσεις για τους νέους οι οποίοι θα μπουν σε κύκλο εκπαιδεύσεων μπορεί να το θεωρήσουν αυτό ως μια εξέλιξη αλλά πιο ηλικιωμένα πρόσωπα θα αντιμετωπίσουν τις χέρειες. Άρα και αυτή η λύση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Έχω μία ε, παρατήρηση να κάνω προκειμένου. Φαίνεται να υπάρχουν υπερβολικά πολλά προγράμματα, υπερβολικά πολλοί στόχοι, ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε στην ουσία τα ίδια δημοσιονομικά μέσα, τα ίδια ταμεία, για διαφορετικούς στόχους. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι λείπει η ορατότητα, δηλαδή δεν είναι σαφές πλέον ποια κονδύλια μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον α ή τον β στόχο. Έχω και μια πλέον συγκεκριμένη ερώτηση να σας θέσω. Πώς συνδέονται τα διάφορα κοινωνικά ευρωπαϊκά ταμεία και το Ταμείο υπέρ του επιχειρήν. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά δεν κατανοώ πώς θα λειτουργήσει. Η τρίτη μου παρατήρηση έχει ως εξής, αν μου επιτρέπετε, αναφέρεται στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Όπως είπε και ο κύριος Όρη προηγουμένως, δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την πρότασή σας. θα έλεγα μάλιστα ότι μας εκπλήσει, διότι υπάρχει αυτή η πολύ γενναιόδορη αγροτική πολιτική που διαθέτει πολλά ε, κονδύλια, πολλά μέσα, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση ή κυρίως για σκοπούς εξυπηρέτησης της αγροτικής πολιτικής. Πρόκειται λοιπόν για μια συγκεχημένη κατάσταση όπου βλέπουμε κονδύλια να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν είναι ούτε συνεκτικοί ούτε ξεκάθαροι. Εξάλλου, η αρχική στόχη του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο. Θα μπουν μοιραία σε δεύτερο πλάνο, διότι δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για να επιτευχθούν αποτελέσματα στους τομείς αυτούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν δεν νομίζω ότι θα ε, ταχθεί υπέρ αυτής της προτάσεώς σας. Είπατε κι εσείς ότι πρέπει να αρθούν τα κολλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά της απασχόλησης, στην ενή αγορά δηλαδή. Ήθελα να σας θέσω την ερώτηση είναι Ολομέλεια, αλλά δεν πρόλαβα. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που θα θέσω την ερώτηση μου αυτή. Το χαρτοφυλάκιό σας έχει την πρόθεση να εξετάσει ποια είναι τα επαγγέλματα εκείνα που ενδιαφέρουν τις χώρες μέλη για να προσφέρουν την πρόσβαση στις αγορές τους ή και την ηθαγένειά τους. Φαίνεται πως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία μπαίνουν ως προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε την κυρία Στάντρουκ και μετά θα έχετε το λόγο κυρία Στάντρουκ. Στην εισαγωγή σας κύριε Επίτροπε αναφερθήκατε και στο πακέτο της απασχόλησης που υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα είχατε πει ότι οι διαμεθοριακές, ε, ε, ε, διαμεθοριακές εταιρικές σχέσεις θα μπουν στο ΙΑΣΕΦ. E εγώ είμαι και εισηγήτρια για θέματα κοινωνικής μεταλλαγής και διαμεθοριακών ε, δραστηριοτήτων και για ορισμένες από αυτές ισχύει ότι αφορούν τέσσερις χώρες. Εκεί βλέπω να υπάρχει πρόβλημα για το μέλλον των εταιρικών αυτών σχέσεων. Δεν βλέπω κάθετα μέτρα να λαμβάνονται καθόλου και όπως είπα φύγονται μέχρι και τέσσερις χώρες αναπερίπτωση. Εγώ το έθεξα, το θέμα αυτό και μου είπαν ότι δεν θα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δηλαδή η διοικητική ε, δράση του προγράμματος να, να, να, καλύψει και τις τέσσερις χώρες. Πώς σκέπτεστε, όλοι θέλουμε την κινητικότητα των απασχολουμένων και την μεγαλύτερη κινητικότητα την έχουμε ακριβώς σε παραμεθόριες περιοχές. Στο μέλλον πώς θα την εξασφαλίσετε αυτή την κινητικότητα. Έρχομαι στην τοποθέτηση πάλι της Ελίζαμπεθ Σρόιντερ για την απόσπαση των εργαζομένων. Οι έλεγχοι, είπατε, θα μειωθούν. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Σρόιντερ. Έχω πάει κατ' επανάληψη και στη Γαλλία και στη Γερμανία σε οικοδομές όπου διαπίστωσαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τον έλεγχο επιχειρήσεων του γραμματοκιβωτίου όπως λέγονται, που δεν είναι πραγματικές εταιρείες δηλαδή. Δεν ξέρουμε πώς να τις ελέγξουμε και με τη συνεργασία με τις ε, τοπικές διοικητικές αρχές. Στις υποχρεώσει του απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση πρέπει πρώτα-πρώτα να ρίξουμε το βάρος. Να εξετάσουμε δηλαδή εάν οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι γνωρίζουν και πού μπορούν να στραφούν και μάλιστα να λάβουν την ενημέρωση αυτή και στη μητρική τους γλώσσα. Ακόμα πιο έντονα είναι τα προβλήματα στις αλυσίδε υπεργολαβιών. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα από την πράξη που μπορώ να διαβιβάσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο από τον τομέα της οικοδομής. Και όλα αυτά μου δείχνουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ελέγχους, δηλαδή και στη χώρα αποστολής και στη χώρα υποδοχής και σε ό,τι, Ευρωπα... και σε ό,τι αφορά τα δίκτυα που λειτουργούν μέσα στην Ευρώπη. Βέβαια κάπου κάπου έχω ανάγκη να επενέσω κιόλας τον Επίτροπο τουλάχιστον για αυτά που είπε για τον ελάχιστο μισθό που ισχύει στην πατρίδα μου τη Γερμανία και για τα οποία είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Από την άλλη μεριά βλέπω όμως και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες εκείνες οι οποίες λαμβάνουν υποστήριξη και όπου εν τέλει παρεμβαίνουν στους κατώτατους μισθούς και στις συμφωνίες που κάνουν οι εταίροι στις συλλογικέ συμβάσεις. Βλέπω δηλαδή εδώ να υπάρχει κάποια αντίφαση, μια σύγκρουση. Θα ήθελα εδώ να μου εξηγήσετε λίγο περισσότερο περί κατώτατων μισθών αλλά και ελάχιστων προδιαγραφών για την απασχόληση. Προκτήθεστε να κάνετε κάτι στο μέλλον. Ε, Κύριε Επίτροπε, απαντήστε πρώτα σε αυτές τις ε, παρεμβάσεις γιατί κάθε μια από αυτές είχε πολλές ερωτήσεις. Μετά Εκτός από αυτούς, άλλοι, η κυρία Ντελή, καλά κλείνω τον κατάλογο των παρεμβαίνοντων. Ο κύριος Επίτροπος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο μέτρο του δυνατού. Ήμουνα αρκετά γρήγορος στους προηγούμενους γύρους για να σας δώσω πιο πολύ χρόνο Πιστεύω το πακέτο του ασχόλησε είναι κατά κύριο λόγο πρακτικό και στην ανακοίνωση για τους τρεις ε, τομείς γίνεται παρκής αναφορά για την χρήση της μαθητείας και πώς η μαθητεία θα πρέπει κανονικά να οδηγεί, ε, να, να οδηγήσει σε μια συμφωνία στο τέλος χρονιάς. Αυτή τη τομή δεν είναι αποκλειστική και μόνο υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες και απλά λέμε ότι υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι θα έχουμε αυξητικές τάσεις για παράδειγμα στον, στην πράσινη οικονομία, θα έχουμε αύξηση των θέσεων εργασία και χρειάζονται όμως κατάλληλες δεξιότητες, επενδύσεις και κατάλληλες πολιτικές για να μπορέσουν πραγματικά να έχουμε περισσότερες εργασίες στην Ευρώπη. Σε καλή συνεργασία βεβαίως με τους συναρμόδιους ε, επιτρόπους, δηλαδή τους επιτρόπους και θέματα περιβάλλοντος, ε, υγείας κτλ. Το Επιτροπό για παράδειγμα. Και στην υλοποίηση βεβαίως χρειάζεται μια συνεργασία μεταξύ όλων των καθήλων αρμόδιων φορέων. Επειδή το κείμενο δεν με τη διατύπωση που επιλέγουμε δεν αποκλεί ούτε αποτρέπει την, ε, τον δεχόμενο περαιτέρω πρωτοβουλειών και νομοθετικών πρωτοβουλειών. Τώρα μιλούμε για μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασία, αυτό κατά κύριο λόγο συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρο στα κράτη-μέλη. Συχνά αυτές οι μεταρρυθμίσεις αφορούν ιδιαίτερες εθνικές πραγματικότητες. Οπότε διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δεν μπορούν λοιπόν να υπάρχει μια ενιαία μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα θα γίνουν πολλές συζητήσει επί του πακέτου μετά δηλαδή με το ε, Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μιλήσουμε στους κοινωνικούς ατέρους στην Επιτροπή Απασχόλησης και το Σεπτέμβρη θα υπάρξει και μια διάσκεψη όπου θα στήσουμε και αναλυτικά πρακτικά ζητήματα αλλά όχι μόνο. Εκεί μπορούν να ακουστούν και άλλες ε, προτάσεις για την καλύτερη υλοποίηση του πακέτου. Σίγουρα λοιπόν δεν τελειώνει εδώ η διαδικασία. Μάλλον αρχίζει μια νέα προσήγηση, μια νέα περίοδος ενασχόλησης με το θέμα και την προσπάθεια της Ένωσης να ξεφύγει από την ύφεση και να οδηγηθεί σε τροχιά ανάπτυξης θέσεων εργασίας. Το EGF τώρα, κυρία Μπάουερ. Το παρουσιάζουμε μία νέα προσέγγιση, δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά ε, ε, είναι μία προσέγγιση, αν θέλετε, που προσπαθεί να συμπεριλάβει πιο πολλούς, ε, αφορά τους εργαζόμενους προστομής, αλλά και τους αγρότες. Αλλά για τους αγρότες είναι περιορισμένο το μερίδιό τους. Για τους μη αγρότες είναι απεριόριστο το μερίδιο στη νέα πρόταση για το EGF. Και ελπίζω αυτή η προσέγγιση να γίνει αποδεκτή εν τέλει. Αλλά αυτό που είπα και νωρίτερα ισχύει και εδώ, αυτό που στη Φραουσέτ. Πρέπει να διατηρήσουμε τη βασική λειτουργία αυτού του εργαλείου, να τη διασφαλίσουμε δηλαδή, να αποκριθούμε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε έκτακτε καταστάσει όπω είναι κλείσιμο επιχειρήσεων ή με την κατάστασή του σε άλλε τρίτε χώρε ή άλλε επίρου. Κάτι που οδηγεί σε ε, ραγδαία αύξηση της ανεργια τοπικά. αυτή είναι η βασική λειτουργία του EGF, να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε απροσδόκητες καταστάσεις. Για τους κατώτατους μισθούς, ναι, ναι, να υπάρχει μια αμφισημία εν προκειμένο και πρακτικά ίσως να φανεί αυτό στις χώρες που είναι στο πρόγραμμα και χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση σε μέγεθος τέτοιο που δεν έχουμε βιώσει, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο καιρό. Ελπίζω η περίπτωση της Ελλάδας να μην είναι παράδειγμα, αλλά είναι εξαίρεση αλλά και η περίπτωση της ε, Ελλάδας που κατάφερε να διασφαλίσει ένα κατά το μισθό, είναι ένα θετικό στοιχείο. Βεβαίω, ε, κατά τι συζητήσει ε, που έγιναν δεν ακούστηκαν. Η άποψη δεν ήταν ενιαία. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Βεβαίω, η συζήτηση με του Έλληνε κοινωνικού εταίρου στην Αθήνα είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και πιστεύω ότι με την περαιτέρω προσαρμογή, την ίδια προσέγγιση θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε σε όλα τα κρατη Όμως, Όμω, το πρόβλημα εμένα αυτή τη στιγμή και κατά κύριο λόγο δεν συνίσταται την ανακολουθία των διαφόρων παραγόντων που θα πρέπει να καθορίσουν το κάτω μισθό, αλλά την εσωτερική υποτίμηση ε, που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές και άρα πώς μπορούμε το κάτω να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της νομισματικής ένασης όταν ε, δεν ε, μπορούμε να μοιραστούμε αν θέλετε τον κίνδυνο. Τώρα για το Μόντι 2 δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων να πω το εξής. Στην πρόταση αυτή φτάσαμε μετά από πάμπολες συζητήσεις. Προσπαθήσαμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία ούτως ώστε να μπορεί να είναι και πρακτικά εφαρμοστέο. Ε, με χαρά λοιπόν να ακούσω και τα δικά σας σχόλια περαιτέρω. Δεν είστε ικανοποιημένοι. Ο Επίτροπος δεν απάντησε δύο από τις ερωτήσεις μου λέει η κυρία Στάνιμπλου, αφενός για τις ε, διαμεθοριακές εταιρικέ σχέσεις και η άλλη ήταν ε, για την απόσπαση των εργαζομένων. Να ακούσουμε πρώτα τους τρεις εναπομένοντες συναδέλφους και αν υπάρχει χρόνος ακόμη ε, να επανέλθετε με τις δύο ερωτήσεις σας. Κρίστενσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα επανέλθω στην ερώτηση του Στίβεν Χιούζ σε σχέση με τον κανονισμό Μόντι 2. Είμαι βέβαιος ότι έγινε η προσπάθεια να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους κανόνες της ενιαίας αγοράς και στα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί ο Επίτροπος ο ίδιος είπε στο Στρασβουργό ότι δεν πρόκειται για προσπάθεια ευρωπαϊκής ρύθμισης του δικαιώματος της απεργίας. Είπατε σήμερα ότι αυτό ισχύει απεριόριστα. Όμως τότε πώς μπορείτε να αναφέρεστε στα ε, δικαστήρια της εργασίας στα ε, πλαίσια της, ε, του κανονισμού Μόντι αφού όπως είπαμε το δικαίωμα της απεργίας υπάρχει είναι απεριόριστο και μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρξει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συλλογικά μέτρα, οι συλλογικέ συμβάσει δηλαδή, είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Γιατί δεν ακούσατε του κοινωνικού εταίρου, που αυτοί είναι αρμόδιοι για να προτείνουν μέτρα για την για το δίκαιο τη απασχόληση. Αυτά που λέτε είναι αντίθετα και με τη Διεθνή Οργάνωση εργασία, αλλά και με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που ερμηνεύουν το δικαίωμα τη απεργία με τρόπο διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι με τον κανονισμό Μόντι 2 τα πράγματα απλώς δυσχεραίνονται. Η λέει η πρόεδρος ο κύριος Φάλμπρ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε πραγματικά ότι η δέσμη μέτρων που μόλις μας παρουσιάσατε θα βοηθήσει. Εγώ δεν το πιστεύω. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερασπίζει τον εαυτό της, την αγορά της ε, κατά των εισαγωγών εμπορευμάτων από μέρη και χώρες ε, με χαμηλά ημερομίσθια, κακή αντιμετώπιση των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Πώς μπορείτε να ζητάτε, ε, ε για ποιο λόγο δεν ζητάτε ε, τελωνιακά τέλη, κατά, τελωνικούς δασμούς κατά αυτών των αγαθών και τέλος πώς θα ε, υπερασπίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους φορολογικούς παράδεισους όσον αφορά τον ελάχιστο μισθό θα ήθελα να πω ότι σε κάθε βήμα στον κοινωνικό τομέα τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να προσέζουν το επιχείρημα της ε, παράδοσης και της ε, επικουρικότητας ε, και έτσι θα συνεχίσει η κατάσταση των, ε, με τα συμφέροντα των συνδικατών και του χαμηλού μισθού ε, στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Ουγγαρία. Ετοιμάζονται νόμοι για περιορισμού αυτού του δικαιώματο. Εμεί, στο Στρασβούργο κριτικάραμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όσο πιο μακρινή είναι η χώρα, τόσο πιο μεγάλη η επίκριση. Τι γίνεται με τα ανθρωπ... Ε, όταν έχουμε πρόβλημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα εντό τη Ευρώπη παραμένουμε σιωπηλοί. Ευχαριστώ κυρία Κάρη Μαντελή και μετά προτείνω μία μικρή ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους μπαίνει στο δρόμο της οικολογικής και κοινωνικής μετάβασης της οικονομίας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συζητήσω για την πράσινη οικονομία, για την οποία λέτε στο εγγραφό σας ναι, πρέπει να επενδύσουμε στον ενεργειακό τομέα, να αναπτύξουμε εκπαίδευση στις πράσινες τεχνολογίες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η οικολογική μετάβαση. Ωστόσο, μου φαίνεται ότι η Επιτροπή δεν καταφέρνει να προτείνει μια λύση για τους λιγότερο ε, εκπαιδευμένους ε, εργαζομένους και για τους ε, εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Η πράσινες θέσεις εργασίες δεν πρέπει να αφήνουν ανθρώπους στο περιθώριο. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε γι' αυτό. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Το δεύτερο, όταν μιλάμε για πράσινες θέσεις απασχόλησης, πρέπει πρώτα απ' όλα να τονίσουμε την ε, σωστή εργασία, τη βελτίωση των συνθήκων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, πρόκειται να υλοποιήσετε ναι ή όχι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τι συνθήκε υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασία. Στη συνέχεια, όσον αφορά την ευελιξία τη εργασία. η Κομισιόν προωθεί την εσωτερική ευελιξία ώστε να αποφευκθούν οι απολύσει, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως λέτε. Προωθείται και αυτό είναι πολύ καλό την επαγγελματική ασφάλεια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι καταδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κόστος των συμβάσεων αορίστου του χρόνου και λέτε ότι οδηγούν σε κατακαιρματισμό τη αγορά εργασία μεταξύ του CDI και του CDD. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ, όμως εγώ ότι εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή για να μεταρρυθμίσουμε τις συμβάσει αορίστου χρόνου. Τέλος, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν επιτέλους αναγνωρίζει ότι η δουλειά δεν επιτρέπει πλέον στους ανθρώπους να ζήσουν ε, ικανοποιητικά, αξιοπρεπώς. Πολύ ωραία λοιπόν που επιβάλλουμε ελάχιστους μισθούς, ε, κατώτατους μισθούς σε μέρη όπου δεν υπήρχαν. Ωστόσο πρέπει αυτοί οι κατώτατοι μισθοί να εξελίσσονται ευέλικτα και χωρίς να ξεχνάμε το αξιοπρεπές επίπεδο ζωής. Δηλαδή υπενθυμίζω ότι πρέπει να διασφαλίζουμε σε κάθε Ευρωπαίο αξιοπρεπή τρόπο διαβίωσης. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο διαφημίζεται τους κατώτατους μισθούς ε, αναδιάφορους τομείς για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά προσέξτε, επειδή εδώ προσθέτεται έναν κίνδυνο, θα υπάρχει επιπλέον ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Τέλος, θα ολοκληρώσω με ένα πολύ σημαντικό ερώτημα στην κοινωνία μας, το ζήτημα των νέων. Μας αναφέρεται κάτι προφανές, το οποίο υποστηρίχθηκε από τη συνάδελφα από την Εμιλή Τυρινέλ, αυτή την ε, πασίγνωστη πλέον διασφάλιση για την νεολαία το 2012 και κυρίως ένα χάρτη για την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εγώ λέω ναι μάλιστα ας προχωρήσουμε αλλά πιο γρήγορα όμως διότι στη συνέχεια θα χρειαστεί και να την επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη. Τρίτη και τελευταία μου ερώτηση λοιπόν είναι πώς θα καταφέρετε να την επιβάλλετε στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Σε αυτή τη φάση εγώ δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες ε, που θα συζητήσουμε για το καθένα από τα στοιχεία αυτού του προγράμματος. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες ε, ε, να επανέλθουμε σε αυτή τη δέσμη μέτρων που αναφέρατε για την απασχόληση όσον αφορά το, την ωφελημότητα και ε, όσον αφορά και το κατώτατο μισθό που αναφέρεται. Ωστόσο θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο έχουμε ήδη αναφέρει σε πολλές ευκαιρίες που πιστεύω ότι δεν ε, βρισκόταν στον δικό σας χάρτη για το πρόγραμμα εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013 είναι το ζήτημα των σχέσεων με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας υπό δύο πτυχές. Ε, πρώτον, όσον αφορά τις προϋποθέσεις επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον νομική υπόσταση, νομική μορφή, θα φανταζόταν κανείς ότι στο μέλλον θα μπορούσε να είναι ε, μέλος ε, αυτοτελές των συνθήκων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Δεύτερον, τι κάνετε όσον αφορά τις, τα κράτη-μέλη που έχουν ε, ελλειπές track record όσον αφορά την συμμετοχή σε τέτοιες συνθήκες. Επίσης, πώς θα ικανοποιήσετε τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας να συμμετέχει στις, ε, τρόικα, στην εκάστοτε τρόικα ε, που παρακολουθεί μία ή την άλλη χώρα. Έχετε 10 λεπτά κύριε Επίτροπε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές και ενδεχομένω θα μπορούσατε να απαντήσετε και στα ζητήματα που η κυρία Σάιντροκ θεωρεί ότι δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση. Έχω κάνει. Yes, let me start by uh, uh, uh, Ξεκινήσω με κάποια πράγματα για να πω ότι δεν τα ξέχασα, απλά τα παράβλαψα. Για το διομεθοριακή διάσταση του ESF και άλλων σχετικών εργαλείων. Όχι, ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις διασυνοριακές δυνατότητες. Το ίδια πρόταση για το Ταμείο κάνει πιο ρητές στιγμένες αναφορές σε σχέση με ό,τι ισχύει στο παρελθόν. αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες, κάποιοι περιττοί για αδικαιολόγητοι περιορισμοί στον κανονισμό για το ESF ή σε κάποιο άλλο εργαλείο, να μου πείτε συγκεκριμένα να το συζητήσουμε. Γιατί φυσικά αυτό αντίκειται στους στόχους. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε όσο γίνεται περισσότερο τη διασυνορική συνεργασία και απασχόληση. Σε ό,τι αφορά τώρα τους λεγόμενους περιορισμούς στην απόσπαση των εργαζομένων και στην πρόταση και τα κλαδικά ζητήματα, τα κράτη-μέλη μπορούν να οικοδομήσουν πάνω στην πρόταση οδηγίας και να ε, νομοθετήσουν περαιτέρω. Είπαμε ότι θα πρέπει και στο κατασκευαστικό κλάδο να ε, να νομοθετήσουν την ρήτρα για την κοινή περιβαλλοντική ε, ευθύνη και αυτό θα πρέπει να μην περιοριστεί σε αυτόν τον κλάδο. Τώρα για τον κανονισμό Μόντι 2. Κατά τι λοιπές του διατάξεις, ο κύριος Κρίστενσεν επέστρεψε στο ίδιο ζήτημα και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα στην απεργία με το άλλο ισχυρό δικαίωμα πάλι του ανθρώπου που είναι ε, η βασική ελευθερία της εγκατάστασης και του επιχειρήν που είναι βασικές αρχές και δικαιώματα που ε, ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την γέννησή της. Εμείς στην πρότασή μας ε, τεκμηριώνουμε πιστεύω επαρκώς την πρότασή μας. Πιστεύω ότι τα δύο στοιχεία άλλως συμπληρώνονται και προσαρμόζονται στην ε, εκάστοτε κατάσταση. Το δικαίωμα, αν θέλετε, στην απεργία είναι μια εγγύηση και είναι η δυνατότητα αντίδρασης του εργαζόμενου στην εξημερινή κατάσταση. Και από την άλλη υπάρχει το θεμελιώδες δικαίωμα στην παροχή υπηρεσιών ή το δικαίωμα στην εγκατάσταση. Και μάλιστα στον κανονισμό Μόντι 2 προβλέπονται συγκεκριμένοι μηχανισμοί που είναι πρακτικά εργαλεία για να αποτρέψουν τη συγκρούση ανάμεσα σε αυτά τα δικαιώματα. Και αυτό έχει φανεί εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό στο παρελθόν. Ο κανονισμός Μόντι 2 λοιπόν προβλέπει καλύτερους τρόπους επίλυσης τέτοιων διαφορών. Τώρα, αυτό το πακέτο, οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία της Κομισιόν θα πρέπει να υπερασπίζεται την μια αγορά καλύτερα. Ήταν ένα άλλο επιχείρημα που ακούστηκε. Θεωρώ ότι αυτή τη δήλωση θα πρέπει να τη δούμε με μεγάλη σύνεση και επιφύλαξη. Και να δούμε αν εδώ έγκαιρε το βασικό πρόβλημα. Αν δούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το εμπορικό συζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δούμε ότι είναι θετικό. Οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα εν προκειμένου στην ε, θέση σε εμπόρια ευρωπαϊκών προϊόντων σε άλλες αγορέ. Οι εμπορικές μας σχέσεις ε, με άλλες χώρες, αν λάβουμε υπόψη τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια κτλ, βλέπουμε ότι ε, το εμπορικό συγγείο είναι θετικό. Όμως πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές όταν βλέπουμε γενικότερα τις οικονομικές μας σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο και να αποφύγουμε τον προστατευτισμό. Η, τα κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική προστασία είναι σημαντικά στοιχεία στα οποία έχουμε επιμείνει στις συμφωνίες που έχουμε με άλλες χώρες του κόσμου ε, είναι θέμα που έχει απασχολήσει το G20 τα τελευταία χρόνια και γίνει σημαντική δουλειά σε αυτό το τομέα και υπήρξαν και πολύ καλά συμπεράσματα για την ε, θέσπιση ενός ελάχιστου επίπεδου κοινωνικών ε, δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού διαλόγου και αυτό λοιπόν υπάρχει και είναι θεσμοθετημένο με τους ε, εταίρους μας τώρα για τις δημόσιες προμήθειες και σε αυτό το τομέα Προσπαθούμε να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Ξέρετε την συγκεκριμένη πρόταση που έκανε ο Επίτροπος Μπαρνιέν προκειμένου. Βεβαίω αναφέρατε πράγματα που είναι χαρτοφυλάκια άλλων ε, επιτρόπων, δηλαδή τα θέματα εμπορίου, η φορολόγηση κτλ. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Αλλά Σίγουρα οι πολιτικές ε, συνάπτονται εφάπτονται και σίγουρα να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων μας. Τώρα, σχετικά με τους εργαζόμενους με τις λιγότερες δεξιότητες και κατά πόσο καλύπτονται αρκετά από το πακέτο προτάσεων. Ναι, είναι κατηγορίες εργαζομένων που έχουμε λάβει υπόψη, όμως και εδώ πάλι θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και ποιο είναι η προσέγγιση να το ακολουθήσουμε. Με του πιο ηλικιωμένου, για παράδειγμα, εργαζόμενου, υπάρχει η Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία για την Ενεργό που ουσιαστικά δεν κάνει μόνο προτάσει, αλλά ε, προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Και μάλιστα στην αγορά εργασία βλέπουμε ότι ακόμα και την περίοδο τη κρίση οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι δεν είναι το πρόβλημα. Βλέπουμε ότι ετησίω αυξάνει ο αριθμό των ε, πλέον ηλικιωμένων εργαζομένων και για τους λιγότερο, ε, τα άτομα με λιγότερες δεξιότητες, ο στόχος είναι να αποκτήσουμε περισσότερε δεξιότητες, Σίγουρα. Αλλά αν δείτε την κατάσταση στην αγορά εργασίας θα δείτε ότι δεν είναι οι εργαζόμενοι με λιγότερες λιγότερε που ε, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Είναι οι μέσε κατηγορίες που έχουν πληγεί περισσότερο. Ξέρετε, είναι το φαινόμενο της πόλωσης αγοράς εργασίας, δηλαδή τη μεγαλύτερη απόλυτη εργασία αφορά τις μεσαίες κατηγορίες εργαζομένων. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε τώρα τις μας προσπάθειες. Φυσικά χρειάζονται προσπάθειες στρατηγικές για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Όταν όμως μιλάμε... Εμ, όταν μιλάμε όμως για προσπάθειες και στρατηγική θα πρέπει να εντοπίσουμε ποια είναι τα προβλήματα και ποια είναι τα πλέον σοβαρά προβλήματα. Κυρία Ντελή, για τα θέματα υγεία και ασφάλεια χορηγασία, συμφωνώ μαζί σα. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μια νέα στρατηγική, όμω πρέπει να γίνει μια πρώτα αξιολόγηση. Είχα την ευκαιρία την προηγουμένη Παρασκευή ε, να λανσάρω μια νέα εκστρατεία για αυτό το θέμα εδώ στις Βρυξέλλες με τον οργανισμό των Bilbao και είχα την ευκαιρία να πω ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ταυτόχρονα να προετοιμάσουμε το περιεχόμενο μιας πιθανή νέα στρατηγική. Αν μπορείτε και σας μα βοηθήσετε για να εντοπίσουμε στοιχεία κλειδιά για μία νέα μακρόπνο ε, στρατηγική θα ήταν ευπρόσδεκτο. Επίσης, το άλλο θέμα που θέσατε θα συζητηθεί αύριο στο άτυπο ΕΨΚΟ, στο Συμβούλιο Προγράμμα που θα λάβει η χώρα στην Δανία. Ναι, ναι, μαζί με την Πρόεδρο θα συζητήσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό των εγγύσεων με τους ίδιους τους υπουργούς και ελπίζω να καταλήξουμε σε πρακτικά συμπεράσματα μέσω αυτή της διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO, ξέρετε, και προσωπικά αλλά και θεσμικά ε, σε συνεχή συνεργασία με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόληση έχουμε ε, δουλέψει πάνω στο θέμα. Π.χ. έχουμε κάνει μια κοινή έρευνα με το ε, ILO για τις πράσινες εργασίες. Είναι κομμάτι του πακέτου απασχόλησης, και το παρουσιάσαμε το περασμένο Νοέμβρη στην Γενέβη με τον Γενικό Γραμματέα του ILO. Και μάλιστα μια ανακοίνωση της Κομισιόν του 2008. Ήδη είχαμε καλέσει και τα κράτη-μέλη να κυρώσουν αυτή τη σύμβαση. Άρα λοιπόν περιμένουμε τώρα την ιδρύση των κρατών μελών. Θα σε ενημερώσω όμως σχετικά για τη διαδικασία εν αυτό το χρόνο. Από εκεί και πέρα, οι υπηρεσίε μα είναι έτοιμε να ξεκινήσουν την εκπόνηση μια μελέτη για το θέμα αυτό. Το... Και τα αποτελέσματα βεβαίω θα τα μοιραστώ μαζί σα όταν θα ολοκληρωθεί η σχετική ανάλυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. obviously... Καλά λοιπόν. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μπει στον διαρθρωμένο διάλογο που θα διεξαγάγουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Αναμένουμε το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε και στην απάντηση του Συμβουλίου. Και σε ό,τι αφορά εμάς, σε διμερή βάση, βεβαίως, αλλά και πολύ σύντομα πάλι και με το σύνολο της Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. <laughs>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 Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ξανακαθίσετε. Σας προτείνω, μην καθυστερούμε γιατί έχουμε πολύ πλούσια ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα. Σας προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας παρότι μόνο οι μισοί ομιλητές μας βρίσκονται εδώ σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ράιμερ Μπέγκε. Σας ευχαριστώ που βρίσκεται μεταξύ μας από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Φυσικά είναι πολύ σημαντική για εμάς αυτή η συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Δημοσιονομικό πλαίσιο για το οποίο όπως γνωρίζετε η Επιτροπή μας θα πρέπει να συντάξει γνωμοδότηση και που σήμερα έχει μπει σε μια καινούργια φάση καθώς το Συμβουλίο Γενικών Υποθέσεων αποφασίζει κομμάτι προς κομμάτι για αυτό που ονομάζουμε το κουτί των διαπραγματεύσεων όπου έλαβαν επαφές μεταξύ των διαφόρων εισηγητών αυτού του κοινοβουλίου, οι οποίοι γεμίζουν μια αίθουσα σαν αυτή είναι εδώ. Αν υπολογίσουμε όλους τους συζητητές όλων των επιτροπών, τόσο για το δημοσιονομικό όσο για το νομοθετικό κομμάτι, όλοι λοιπόν εξέφρασαν κάποια ανησυχία όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο, ανεξάρτητα από την ταχύτητα των δικών μας εργασιών. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συνεδρίαση ε, γίνεται σε αυτή την ειδικά επιλεγμένη στιγμή. χωρί λοιπόν καθυστέρηση δίνω το λόγο στον κύριο Μπέγκε για να μας παρουσιάσει το στάδιο του προβληματισμού και των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Από την άποψη της πολιτικής συνοχής, ε, αυτή θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της αυριανής ημέρας. Όπως γνωρίζετε όλοι, δεν είναι μυστικό, η παρούσα Επιτροπή έχει ζητήσει μια ε, διαδικασία συνδεδεμένης επιτροπής σε αυτό το τομέα δεν θα το συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, αλλά ανήκει αυτή η πρόταση σε αυτό το τοπίο όπου αυτή η Επιτροπή θεωρεί ότι στο πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απασχόληση, όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις στο κάθε κράτος μέλος, τόσο λόγω της κρίσης αλλά και όσον αφορά τα σχέδια ε, εξυγίανση των δημοσιονομικών οικονομικών η παρούσα επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχει σημαντικά στον ορισμό των όρων επέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων διότι ε, αν δείτε τι περιλαμβάνεται σε αυτό το γενικό πλαίσιο πρώτα απ' όλα υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ρητά ορισμένα ταμεία τρία ταμεία το, το Ταμείο Περιφερειακής Συνεργασίας το διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας ή των ενδιάμεσων περιφερειών. Είναι θέματα που αφορούν άμεσα τις προϋποθέσεις επέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν συζητώ λοιπόν να υποστηρίξετε το ένα ή το άλλο να ασκήσετε κάποια λειτουργία που δεν είναι η δική σας, αλλά θέλω να περιγράψουμε το γενικό πλαίσιο παρέμβασης μας στο πλαίσιο της παρουσίας Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πνεύμα και να έχουμε το πνεύμα αυτό τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε αυτές τις συζητήσεις, δεδομένου ότι έχουμε εντάξει τη διαιτησία που έχει γίνει όσον αφορά τους αριθμούς και ότι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά στην ώρα της ψηφοφορίας δεν θα πρέπει να παρουσιάσουμε νούμερα τα οποία θα προεξοφλήσουν ε, τα δημοσιονομικά πέραν των όσων έχουν αποφασίσει, έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο όταν ενέκρινε την έκθεση της Επιτροπής. Κύριε Σίγητη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε λέει ο κ. Μπέγκε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κανονικά θα έπρεπε να είναι παρόν και ο κ. Καλφίν, που είναι συνεισηγητή για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι όμω και έτσι θα αρχίσω ευθύ αμέσω. Γνωρίζετε βέβαια ότι στην βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα μπαίνουμε πλέον σε μια τελείω διαφορετική κατάσταση από ότι ήμασταν ε, στι συζητήσει για το προηγούμενο Πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το νυν πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να εγκριθεί ομόφωνα από το ε, Συμβούλιο μόνο εφόσον έχει εγκρίνει πρώτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία. Και υπενθυμίζω ότι στι διαπραγματεύσεις για την συνέλευση, για την ε, σύνταξη της ε, συνθήκης τότε, το Κοινοβούλιο επέτυχε την συναπόφαση για τα δημοσιονομικά πλαίσια με συντονισμένη ενέργεια των εθνικών διπλωματών στο άθρο 312 όπου αναλαμβάνουν όλα τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν και να πράξουν πάντο δυνατό ώστε οι διαδικασίες να μπορούν να κινούνται ταχαίως και με συνέπεια. Ακριβώς αυτό εξαργυρώνουμε τώρα και χάρη ε, στην δέσμευση της Πολωνικής και Ουγγρικής Προεδρίας αλλά και στην Ιδανική Προεδρία η διαπραγματευτική ομάδα πενταμελής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την προεδρία του κ. Λαμασούρ, πρόεδρου της Επιτροπής Προπολογισμών, μαζί με τους κ. Ντεχάνε, Αν Γένσεν ως συνεισηγήτρια για τους ιδίους πόρους, συναντώμεθα πριν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για briefing και μετά για debriefing μαζί με τις ε, τρεις προεδρίες. Και έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση από τη Δανική Προεδρία ότι αυτή η διαπραγματευτική ομάδα η οποία είχε ήδη συναντηθεί όπως ε, έγινε και με την Πολωνική Προεδρία θα προσκληθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την περαιτέρω κίνηση των καλαθιών των διαπραγματεύσεων ε, για τον Ιούνιο. Θα γνωρίζετε επίσης ότι ως Κοινοβούλιο Τούτη τη φορά έχουμε και μια πρεμιέρα, δηλαδή πριν να κάνει τι προτάσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί με την Επιτροπή μας ΣΟΥΡΕ διατυπώσαμε τη διαπραγματευτική μας θέση, την εγκρίναμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην ολομέλειά μας και αυτή η διαπραγματευτική εντολή εξακολουθεί να ισχύει. Και εδώ ισχύει και η δήλωση ότι καταρχήν, και εμείς θεωρούμε ότι είναι μετριοπαθές το αίτημα μας αυτό, εν ώψη μάλιστα της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσεως. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν στις απαιτήσει της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, οφείλουμε να έχουμε 5% παραπάνω από τα κονδύλια του 2013. Και αν δεν είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη, τότε να καθορίσουν τις αρνητικές προτεραιότητες οι οποίες εν τέλει θα εκπέσουν από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Το ακούμε ξανά και ξανά από τις χώρες μέλη, μιλούν για την Ατζέντα 2020 ως βασικό προσανατολισμό και για τη μελλοντική δημοσιονομική πολιτική, το ίδιο επίσης για την έρευνα και την ανάπτυξη, 3% το ΑΕΠ. Μας λείπουν για όλη την Ευρώπη 130 δις ευρώ, σχεδόν ένας ολόκληρος δηλαδή ευρωπαϊκός προπολογισμό στην πολιτική αναπτύξεως 0,7% δεν τα βρίσκω αυτά πουθενά ούτε στους προϋπολογισμούς ε, των χωρών μελών ούτε της Ένωσης με εξαίρεση τρεις-τέσσερις χώρες άρα λοιπόν λείπει κάποια ειλικρίνη εδώ και το τρίτο είναι ότι χρειάζεται να εκτελέσουμε ορισμένα καθήκοντα που εκκρίνουν από τον προϋπολογισμό ότι δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο πλεόνασμα πληρωμών το λεγόμενο, το λεγόμενο rest aliquide διότι μόνο έτσι μπορούμε να διαπραγματευτούμε λογικά και να συζητήσουμε, λαμβάνοντα και αυτέ υπόψη. Και εδώ θα πω ότι εάν 8 χώρες μέλη είπαν, όπως φαίνεται στο Συμβούλιο, ότι θέλουν, θέλουν να καταργήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, αυτό αντιβαίνει ασφαλώς στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα εκπλησόμεθα ξανά και ξανά, διότι για την κινητοποίηση του Ταμείο παγκοσμιοποίηση, τα προηγούμενα χρόνια τα διαθέσιμα κονδύλια, και αυτή είναι η βασική αρχή, δηλαδή να λαμβάνει το Ταμείο αυτό από άλλα τμήματα του προπολογισμού μη διατεθειμένα κονδύλια και πάντοτε τα κονδύλια για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης ήρθαν από διαθέσιμα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο οφείλουμε να επεξεργαστούμε, διότι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να λειτουργήσουν σωστά οι εκροές των κονδυλίων και να κατευθυνθούν σωστά. Εξάλλου, μετά από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διάσκεψη κορυφής των αρχών Μαρτίου, να γίνουν περισσότερα δηλαδή πράγματα για τι μικρές και μεσαίε επιχειρήσει, περισσότερα πράγματα υπέρ τη απασχόληση των νέων, πάλι 8 χώρο μέλη επανεπεξεργάζονται τα επιχειρησιακά τους προγράμματα με αυτούς τους στόχους. Αυτό είναι σωστό. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά για το νομοθετικό υπόβαθρο, για τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις για τα έτη μετά το 2014. Και εδώ θα δηλώσω το εξή. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι στην εξέλιξη αυτή των διαπραγματευτικών καλαθιών ούτε μπορεί κανείς να υποχρεώσει το Συμβούλιο να αναπτύξει κάποιες θέσεις, αλλά πρέπει να έχει μια θέση αν φόσον θέλει να έρθει να μας συναντήσει για τα 65 πολιετή προγράμματα. Αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα το βράδυ με προεδρία του Προέδρου Σούλτς, δηλαδή πώς θα κινηθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πρέπει να είναι σαφές ότι η συζήτηση αυτή για την προώθηση αυτών των διαπραγματευτικών καλαθιών, κουτιών, δεν μπορεί να καταλήξει στο Συμβούλιο Υπουργών στο, ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Αυτά πρέπει να περάσουν πρώτα από τα ειδικά συμβούλια υπουργών. Όχι να πάει κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αρχικών Κυβερνήσεων. Πρέπει να προχωρήσει πρώτα από τα επιμέρους συμβούλια υπουργών. Και αυτά θα παρακολουθήσουμε και εμείς και τα όσα θα ακούσουμε αύριο και τι θα κάνουμε. Αν δηλαδή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιδράσουμε πριν ή μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης εδώ εντάσσεται, όπως είπατε και εσείς μόλις πριν κυρία Πρόεδρε, ότι έχουμε την πρόθεση κατά πάσα πιθανότητα αρχάς Νοεμβρίου να υποβάλουμε ενδιάμεση έκθεση με τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών εν αναμονή κιόλα των μηνυμάτων που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα αποτελέσει λοιπόν αυτή η έκθεση μια ενδιάμεση εκθέση, όπως είπα, βασισμένη στις εκθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, που θα διαμορφώσει την τελική θέση του Κοινοβουλίου για τον τελευταίο αυτό γύρο. Θα είναι λοιπόν μια παράλληλη εργασία που αφενός θα περιλαμβάνει μια προσπάθεια προώθησης των διαφόρων πολιετών προγραμμάτων, όπως είπε και η Πρόεδρος σας προηγουμένως, αλλά ταυτόχρονα και μια γνωμοδότηση, να συνταχθεί μάλλον μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αυτές οι εργασίες μπορούν να αρχίσουν ήδη. Οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών θα πρέπει να είναι έτοιμες το Σεπτέμβριο και να απηχούν και αυτά που θα μας έχει υποβάλει το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι εν ώψη της αμφιλεγόμενης κατάστασης που έχουμε σήμερα στο Συμβούλιο υπάρχουν οι φίλοι της συνοχής, οι φίλοι της αγροτικής οικονομίας και οι φίλοι της αρχής δεν πληρώνω τίποτα με περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ορισμένοι μιλούν για το ποσοστό του ΑΕΠ, άλλοι λένε 100 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Ό,τι και αν συμβάνει αυτό. Ότι αυτοί λοιπόν θα προβούν σε περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και ας μην λησμονούμε ότι παλαιότερα είχαμε φτάσει σε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της τάξης του 1,18% των ε, εσόδων, του ΑΕΠ δηλαδή, Και εδώ πρέπει να μπει και το κέριο μήνυμα της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, όπου η εντολή που μας δίνει είναι η διαπραγματευτική μας εντολή και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε καθαρά στο Συμβούλιο ότι σε περίπτωση όπου δεν συμφωνήσουν δεν θα μπούμε σε κρίση, δημοσιονομική κρίση, διότι τα ανώτατα όρια του περσινού έτους της του τρέχοντος σχεδιασμού παραμένουν ενισχύει μέχρι ότου εξευρεθεί η λύση. Άρα δεν πέφτουμε έξω από το δίκτυο ασφαλείας. Θα υπάρχει ένας προβληματισμός βέβαια σχετικά με την νομική βάση. Αλλά ίσως αυτή η προειδοποίηση και μόνο να αρκέσει ώστε να αντιληφθούν ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Διότι αν εγκριθούν με υπερβολική καθυστέρηση τα προγράμματα και εκτελεστούν στις χώρες μέλη με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και στην πολιτική πολιτική και βέβαια για το 2013. Πάντως εμείς αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια λογική πρόσφορα, μια λογική πρόταση, διότι εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι να καταλήξουμε στην ονομέλεια με μια γνωμοδότησή μας, μια εκθεσή μας δηλαδή, που να λέει ναι ή όχι. Γι' αυτό θα συζητήσουμε με την Προεδρία του Συμβουλίου, θα καταστήσουμε σαφή τη θέση μας και θα εξηγήσουμε ότι όσο πιο δύσκολοι γίνονται οι αριθμοί, τόσο περισσότερη ευκαμψία χρειαζόμαστε για τον πολίτη σχεδιασμό, καθώς επίσης χρειαζόμαστε σημαντικές προόδους στο θέμα των ιδίων πόρων. Επίσης, εμείς ως Κοινοβούλιο σεβόμαστε τη συνθήκη. Οι χώρες μέλη οι οποίες απορρίπτουν τη συζήτηση αυτή φαίνεται να μην έχουν διαβάσει καν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ενώ η συζήτηση περί ιδιών πόρων στο μεταξύ είναι απαραίτητη όχι μόνο για τους ιδιούς πόρους που μας το επιβάλλει η Συνδίκη Λισαβόνας, αλλά και διότι στη συζήτηση περί ιδιών πόρων εκεί απηχούνται όλες οι απόψεις και όλες οι δυσαρέσκειες και επικρίες σχετικά με τους ίδιους πόρους. Νομίζω αυτά πρέπει να έχουν διευκρινιστεί στην αρχή της συζητήσεως τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ. Κύριε Καλφίν, εσεί ευτυχώ μπορέσατε και ήρθατε. Πέστε λίγα λόγια αν θέλετε πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ το συγγνώμη που καθυστέρησα. Χρειάστηκε να προσθέσω μια εκθέση σε μια άλλη επιτροπή. Και έτσι καθυστέρησα. Θα ήθελα να κάνω μερικές συμπληρώσεις ε, για όσα είπε ο κύριος Μπέγκε για το περιεχόμενο του πελετού δημοσιονομικού πλαισίου και θα ήθελα να φέρω και κάποια ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες εντός των επιτροπών. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αύριο θα έχουμε το πρώτο Γενικό Συμβούλιο που θα συζητήσει το υπόλοιπο κομμάτι, το κουτιού διαπραγματεύσεων από την Προεδρία. Το Μάιο θα δούμε ένα σχέδιο του κουτιού διαπραγματεύσεων και τον Ιούνιο η Προεδρία θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υιοθετήσει θέσεις. Βλέπουμε σε αυτό έναν κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε δύο διαδικασίες αντιμετώπισης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου σε σχέση με το Συμβούλιο. Το πρώτο είναι το ίδιο το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, τα νούμερα δηλαδή, και έχουμε τι διαδικασία συνένεση Πρέπει να πούμε στο τέλος ναι ή όχι. Αλλά έχουμε και άλλη μια διαδικασία που αφορά τη νομική βάση και εκεί έχουμε 65 έγγραφα ε, και στην Επιτροπή Απασχόλησης αυτά τα έγγραφα αποτελούν τη νομική βάση και σε αυτά περιγράφονται όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται και, και, και έχουμε την συναπόφαση. Δεν θα είναι λοιπόν αποδεκτό για το Κοινοβούλιο να του στερηθούν τα δικαιώματα συζήτηση ε, για τη συναπόφαση εφόσον ε, οι αρχηγοί κυβερνήσεων αποφασίσουν να δώσουν μια συγκεκριμένη εντολή. Αυτό που εννοώ είναι ότι αν τον Ιούνιο πούν κάτι οι επικεφαλής των κυβερνήσεων, τότε οι υπουργοί είναι πιθανόν να μην το ανοίξουν για διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να προλάβουμε. Θα γίνει μια συνεδρίαση της ομάδας ε, αύριο, στην οποία θα παραστάτε ο πρόεδρος Εκεί πιστεύω θα πρέπει να μελετήσουμε πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου να έχει την ευκαιρία σωστών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για οτιδήποτε θέλουμε να διαπραγματευτούμε. Το δεύτερο κομμάτι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζω ότι το Συμβούλιο δεν ε, θέλει ιδιαίτερα να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει. Ε, ωστόσο, εμεί πρέπει να ξεκινήσουμε, πιστεύω, τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό. Μόλι θα έχουμε μια διαπραγματευτική θέση, για αυτά τα έγγραφα που αποτελούν την νομική βάση. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε θεσμική πίεση στο Συμβούλιο ώστε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις και να συμμετέχει σε αυτό. Σε αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι μια κατάσταση όπου θα λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις από τους αρχικού κυβερνήσεων. Το Συμβούλιο δεν θα έχει διαπραγματευτεί επί της ουσίας με το Κοινοβούλιο και εμείς θα έχουμε ελάχιστο περιθώριο συζήτησης. Όσο λοιπόν το συντομότερο ξεκινήσουμε τις συζητήσεις επί της ουσίας με το Συμβούλιο, τόσο περισσότερες δυνατότητες θα έχει το Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο. Ένα τελευταίο πράγμα, όταν μιλάμε για προπολογισμό, για δημοσιονομικά, όλοι σκέφτονται νούμερα. Και αυτό φυσικά είναι φυσιολογικό. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε να κάνουμε τομιακές συμφωνίες διαφόρων τύπων δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν ας πούμε για το μέγεθος του κονδυλίου, της αγροτικής πολιτικής ή της πολιτικής συνοχής ή για συγκεκριμένα μέσα, μηχανισμούς, αυτό πρέπει να το αποφύγουμε εάν θέλουμε να έχουμε μια ισχύρη διαπραγματευτική θέση με το Συμβούλιο. Η αρχή του ότι δεν συμφωνούμε για τίποτα αν δεν συμφωνήσουμε για όλα θα πρέπει να είναι παρούσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μην μελετήσουν οι επιτροπές τα νούμερα γιατί έχουμε την έκθεση ΣΟΥΡ για παράδειγμα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ρητή αλλά μας δίνει μια γενική εικόνα των μεγεθών και έχουμε και την πρόταση της ε, Κομισιόν. Θα θέλαμε λοιπόν και αυτό είναι δυνατόν ε, να συζητηθεί όλα όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση ΣΟΡ, που αποτελεί εντολή για όλους, για την διαπραγματευτική ομάδα, για την έναρξη διαπραγματεύσεων στις επιτροπές και ούτω καθεξής, πριν η Ολομέλη αποφασίσει κάτι άλλο. Το να μην συμφωνήσουμε λοιπόν στα νούμερα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε για νούμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την κινητοποίηση Ευχαριστούμε που κατά κάποιο τρόπο σε επίπεδο κοινοβούλιο κάνετε αυτό που κατηγορούμε το Συμβούλιο, για, το οποίο... την απουσία του οποίου κατηγορούμε το Συμβούλιο. Να ξέρετε ότι σε αυτή την Επιτροπή θα έχετε συνομιλητές οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να παίξουν συλλογικό παιχνίδι. Δηλαδή θα τηρούν αυτή τη γενική κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τα νούμερα αν δεν συμφωνήσουμε για τα πάντα και ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια στρατηγική στο πλαίσιο της οποίας δεν θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που προχωρούν πιο γρήγορα από άλλους. Θέλουμε να λάβουμε αποφάσεις ως θεσμικό όργανο, είτε σε επίπεδο προεδρίας, είτε σε επίπεδο επιτροπής προπολογισμού, είτε σε επίπεδο ομάδων επαφής και ούτω καθεξής. Κανείς δεν πρέπει να κινείται μόνος του. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα όπως αυτά που αναφέρουμε σήμερα, η συνοχή αφορά πολλές επιτροπές. Εκ μέρους των συναδέλφων και πάλι σας ευχαριστώ για την, για την παρουσία σας, ε, διότι έτσι μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα Αναφέρατε, κύριε Μπέγκε, το ζήτημα του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ότι μέχρι σήμερα αποτελούσε ένα συγκεκριμένο κονδύλιο που τροφοδοτεί από τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εγώ είδα έγγραφα στο πλαίσιο του κουτιού διαπραγματεύσεων τα οποία δεν έμοιαζαν με κουτί διαπραγματεύσεων. Ουσιαστικά μας έλεγαν θέλετε το EGF ή δεν το θέλετε. Θέλετε να αυξηθεί. Είναι εξωφρενικό. Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο απότομη, αλλά πιστεύω ότι επικονίζει την ηθελημένη σύγχυση που διατηρεί το Συμβούλιο η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε καταβαράθρωση των βάσεων στις συζήτησης για το νομοθετικό ζήτημα. Η κυρία Μαρκίν δεν είναι μέσα δαξί μας, αλλά φαντάζομαι ότι ως ε, νομοθέτης ε, για το βασικό κείμενο, όταν εγώ είδα αυτό το κείμενο, αυτό το, αυτές τις ερωταπαντήσεις για τρία σημεία όσον αφορά το μέλλον του EGF ε, στο Συμβούλιο αναρωτήθηκα για ποιο λόγο ε, κάνουμε όλη αυτή την ε, μελέτη και όλη αυτή την άσκηση. Ε, είπατε ότι ε, εν τέλει αν δεν συμφωνήσουμε για τίποτα μέχρι το τέλος του έτους θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε κάτι προσωρινό. Εγώ τι θα κάνουμε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει τη μάχη με το Συμβούλιο και τελικά η κυρία Μέρκελ θα τηλεφωνήσει τον κύριο Μπλερ και δεν ξέρω σε ποιον και όλοι θα πρέπει να σιωπήσουμε Δυστυχώς ή ευτυχώς ε, έχουμε ξαναζήσει δύο φορές αυτού του τύπου τη διαδικασία. Μου έχει συμβεί να εκπλαγώ για το πώς υποχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα διατησίας που δεν έλαβε καν χώρα στις Βρυξέλλες ε, αλλά στη μία ή την άλλη πρωτεύουσα ε, Μπορείτε να φανταστείτε γιατί μιλάω. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ε, στην παρούσα φάση το Κοινοβούλιο πραγματικά αρχίζει να ε, καταδεικνύει την ισχυρή του βούληση να συμμετέχει στις συζητήσεις. Μου φαίνεται ότι αυτή τη φορά ε, τα πράγματα είναι κάπως ιδιαίτερα όπου η πιθανή ένταση μεταξύ της αξιολόγησης του προπολογισμού και εθνικών στρατηγικών υπάρχει κίνδυνος να είναι πολύ έντονη. Το τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω για να σας ε, αναφέρω ουσιαστικά τους δισταγμούς, τις ανησυχίες, τους ενδιασμούς αυτής της ε, Επιτροπής σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο που έχετε να μελετήσετε. Ανέφερα προηγουμένως το ζήτημα της δυναμικής μεταξύ των διαφόρων επιτροπών, αλλά αυτό ήταν απλά για να σας το υπενθυμίσω. Αλλά ήθελα να σας προειδοποιήσω για ένα πρόβλημα πέραν του κατά πόσο το κουτί διαπραγματεύσεων προεξοφλεί τα εργαλεία νομικής βάσης πέραν των νομικών βάσεων ο τρόπος με τον οποίο ήδη προβλέπει τα αποτελέσματα των νομικών βάσεων η Κομισιόν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, τα διαρθρωτικά ταμεία για τα οποία την πολιτική συνοχή για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θέσει ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο δεν θα συζητηθεί πουθενά και το οποίο κυκλοφορεί ήδη σαν να έχει αποφασιστεί. Βρισκόμαστε λοιπόν ε, μεταξύ σφύρας και Ακμωνοστό, στο ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν, ε, της Κομισιόν που μας δίνει οδηγίες χρήσης πριν να έχει μελετηθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε αυτή τη διπλή τάση για τους ε, διαπραγματευτές σε δημοσιονομικά θέματα. Ε, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά θεώρησα ότι θα είναι σημαντικό να αναφερθώ σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ε, κύριε Λόπες, ποιοι άλλοι συναδέλφοι θα ήθελαν να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κυρία Σρέντερ, όχι. Αλήθεια. Κύριε Κούντς. Και ο κύριος Σέρκας. Κύριε Σρέντερ, για το ΕΛΚ η κυρία Μπάουερ. Κλείνει ο κατάλογος. Ε, κυρία Κούντσα. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως μαθαίνουμε είναι περίπλοκη η διαδικασία. Αφενός είναι οι ειδικέ επιτροπές που διαπραγματεύονται επιμέρους ε, θέματα και στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών έχουμε αρχίσει, από εκεί έρχομαι τώρα, έχουμε αρχίσει με αυτούς τους προκαταρκτικούς τριμερείς διαλόγους. Το Συμβούλιο φαίνεται να είναι ανοιχτό για το θέμα αυτό. Βέβαια δεν είναι από τα πιο δύσκολα θέματα αυτός ο φάκελος. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το μείζον πρόβλημα έγκυται ή εντοπίζεται περισσότερο στη διαδικασία για το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και επίσης ε, εκεί τα νούμερα πόσο μεγάλα είναι. Δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα από την αρχή. Θα ήθελα όμως να σας ερωτήσω εάν θα είναι χρήσιμο να καταλήξουμε σε κάποιο ψήφισμα ή κάτι άλλο ώστε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα. Δηλαδή τι αναμένουμε από το Συμβούλιο, τι αναμένουμε να δούμε, πώς να διεξαχθεί η διαδικασία. Να είναι μια ταυτόχρονη παράλληλη διαδικασία που θα εργαζόμαστε επί διαφόρων φακέλων ταυτόχρονα. Αλλά εδώ βλέπω κάποιους κινδύνους αφενός να μην υπάρξει θέση του Συμβουλίου, να μην έχουμε δηλαδή το Συμβούλιο ως εταίρο μας για να ξεκινήσουμε τριμερή διάλογο. Και ο άλλος κίνδυνο είναι να υπάρξει πρόωρος, ε, ε, ε, συνένεση στο Συμβούλιο απόλυτα ξεκαθαρή για αυτούς και να μην μπορέσουμε να την τροποποιήσουμε. Γι' αυτό ίσως πρέπει να διαπραγματευτούμε και την διαδικασία. Να είναι δηλαδή αρκετά εύκαμπτη, ευέλικτη, να μπορεί να λάβει υπόψη και τις γνωμοδοτήσεις των επιμέρους επιτροπών, αλλά βέβαια και το θέμα του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή αυτό, αλλά βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε στην αρχή την διαδικασία. Πώς θέλουμε, πώς θέλουμε δηλαδή, με ποιο τρόπο θέλουμε δηλαδή να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι για τη σοσιαλιστική ομάδα είναι πολύ σημαντικό να μην παραγνωρίζουμε την, την παρατήρηση που κάνατε εσείς, Πρόεδρε, ότι αυτή η διαπραγμάτευση είναι μια συλλογική διαδικασία. Να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι βλέπουμε μπροστά μας και είμαστε μάρτυρες μια πρώτης θεσμικής, αν θέλετε, συζήτηση μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνα. Και εκεί, αν θέλετε, θα δοκιμάσουμε και τις αντοχές της Συνθήκης. Το Συμβούλιο τι κάνει. Καταφέρνει να κάνει το Κοινοβούλιο έναν απλό παρατηρητή για μια σειρά πολιτικών, κυρίως είναι πολιτικές που είναι εικόνα της Ένωσης στον ε, κόσμο. Σίγουρα, αυτό που είπατε Πρόεδρε θα πρέπει να μην το ξεχάσουμε, ότι είναι μια συλλογική μάχη αυτή την οποία δίνουμε. Θα πρέπει το Συμβούλιο να βλέπει επιτέλους το Κοινοβούλιο ως ισότιμο νομοθέτη. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να επισημάνω και είναι σημαντικό να πω ότι είναι κόκκινη γραμμή για τους σοσιαλιστές. Και θα πρέπει να κρούει ο κόδωνας του κινδύνου κάθε φορά που προσπαθεί να περάσει αυτή η κόκκινη γραμμή το Συμβούλιο. Τι εννοώ, όπως είπε ο κύριος ε, Καλφίν και ο κύριος Μπέρκε, παρά τα αυτά, ε, ε, εγώ βλέπω ότι κάποια κρατημέλη, κάποιοι υπουργοί, κάποιοι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν ότι υπέγραψαν τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να τηρούμε αυτά που έχουμε υπογράψει. Και η στρατηγική του 2020 εμπεριέχεται σε συνθήκες και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Το Συμβούλιο έχει συνυπογράψει αυτές τις συνθήκες. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή την οποία θέτει η σοσιαλιστική ομάδα. Υπάρχει μία σειρά κοινών πολιτικών που θα πρέπει να πρικίσουμε οικονομικά. Ιδάλλως όλα θα μείνουν στα λόγια η Επιτροπή Απασχόλησης, η ομάδα μας τουλάχιστον, να πω ότι θα σας υποστηρίξει στο έργο σας, γιατί είναι μίζωνος ε, συμφέροντος να ακουστεί ξεκάθαρα και πολύ χειρά η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς υπερασπίζεται την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή κοινωνία σε μια εποχή ε, κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ε, Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έχω την αίσθηση ότι ετέθη το βασικό ερώτημα από τους προλαλήσατες, ιδίως από την κυρία Πέρες. Εγώ να προσθέσω μόνο κάποια επιμέρους ερωτήματα για το EGF. Ποια είναι η θέση σας σε ό,τι αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε σχέση με τον προπολογισμό. Δεν γνωρίζω κατά πόσον προσπαθείτε να δείτε συνεκτικά, αν θέλετε, τις διάφορες πολιτικές κατά διάφορα εργαλεία. Γιατί εδώ στην Επιτροπή μας αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με την ε, εν μέρη προσχώρηση της αγροτικής πολιτικής στο EGF. Δεν ξέρω κατά πόσον δηλαδή μέσα στην εμβέλεια του ενδιαφέροντός σας είναι και αυτό το θέμα ή όχι. Αν ναι, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Δύο θέματα. Πρώτο, το γεγονός ότι η παρούσα Επιτροπή φέρει την ευθύνη για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που πολύ συχνά πάνε να το κόψουν ως κονδύλι οι χώρες μέλη. Το εργαλείο δηλαδή που ως τώρα λεγόταν Progress και τώρα λέγεται PSCI που είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ενεργαλείο, μάλλον για πιλωτικά προγράμματα σε πολλούς τομείς. Αυτό κινδυνεύει πάντοτε να πέσει θύμα της μάχερας των χωρών μελών. Ως Επιτροπή εμείς προβληματιζόμαστε εάν το εργαλείο αυτό το εξοπλίσουμε με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ως έξτρα προστίκη. Το τμήμα δηλαδή που προτείνουμε εμείς μέσα στην αύξηση δηλαδή του προπολογισμού και με αυτό. Για μένα αυτό σημαντικό είναι πρώτον τι ρόλο παίζει το εργαλείο αυτό στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις και στην προπαρασκευή των διαπραγματεύσεων είναι από τα λίγα και σημαντικά εργαλεία κοινωνικών πιλωτικών προγραμμάτων πού μπορεί να εκπληρώσει τις αιτήσει μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερο, αν θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να συζητήσουμε την δική μας πρόταση για την αύξηση του εργαλείου αυτού. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα αναφέρεται σε ένα θέμα, δεν ξέρω δηλαδή αν μπαίνει αυτό όμως τα θέματα του MFF. Το ερώτημα δηλαδή αν τα κοινωνικά ταμεία μπαίνουν μέσα στη μακροοικονομική επιφύλαξη. Δηλαδή, αν ε, εμπίπτουν δηλαδή στη μακροοικονομική επιφύλαξη. Αν δηλαδή μια χώρα μέλος έχει χρέη, τότε δεν λαμβάνει ευρωπαϊκά χρήματα και αυτό αφορά και τα διαρθρωτικά ταμεία. Που ωστόσο τα διαρθρωτικά ταμεία σε περίπτωση που μια χώρα βρίσκεται σε κρίση είναι και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να βοηθηθεί να ξεφύγει. Δηλαδή πρόκειται για πραγματικές επενδύσεις που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει να ξεπεραστεί η κρίση. Πρόκειται για μια αντίφαση λοιπόν εδώ. Δηλαδή πάμε, μας ζητάνε να κόψουμε, ακριβώς, περικόψουμε εκεί ακριβώς όπου είναι και η μόνη δυνατότητα για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια χώρα από την κρίση. Διαρωτώ είναι και αυτό το τμήμα της διαπραγμάτευσης, αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Και δεύτερο, εάν αποτελεί τμήμα των διαπραγματεύσεων, ποια είναι η θέση της διαπραγματευτικής ομάδας επ' αυτού. με την ίδια σειρά. Πρώτα ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας. Το θέμα της διαδικασίας και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες εξελίξεις για τα διαπραγματευτικά καλάθια και τα σχετικά έγγραφα και πώς θα προχωρήσουμε με το Συμβούλιο. Αυτό ασφαλώ θα παίξει ένα ρόλο στι συζητήσει τη διαπραγματευτική ομάδα. Δηλαδή, ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το ζήτημα λοιπόν θα δώσουμε μηνύματα, θα διευκρινίσουμε ότι εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα όπου υπερβαίνουν κάποιες, κάποια όρια δικά μας, κάποιες λεγόμενες ερυθές γραμμές, δεν θα ε, συμφωνήσουμε, δεν θα προχωρήσουμε. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία να είναι πράγματι πάρα πολύ εύκαμπτη, γιατί κανείς από εμά δεν γνωρίζει μέχρι πού θα φτάσει στα διαπραγματευτικά αυτά καλάθια η ιδανική προεδρία. Δεν θέλω να βάλω νούμερα. Αν όμως υπάρχουν κάποιες βασικές συμφωνίες που θα αποτελέσουν τον πυρήνα και τη διαπραγματευτική διαδικασία για τα μεγάλα προγράμματα, για τη συνοχή, για την αγροτική πολιτική, για την έρευνα, τότε μπαίνουμε πλέον στην ουσία της διαδικασίας συναπόφασης. και ελπίζουμε τότε το Συμβούλιο να καθίσει να σκεφτεί την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την Ατζέντα 2020, διότι θα έχει τότε και θέση για να μπορέσει να διαπραγματευτεί μαζί μας. Το πρόβλημα όμως είναι, εάν αυτά αρθούν σε επίπεδο κάποιων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τότε οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις θα φέρουν ήδη το βάρος αυτών των αποφάσεων. Θα είναι προεπιβαρημένες, αν μπορώ να το πω έτσι σε κάποια χρονική στιγμή θα χρειαστούμε όλοι πολύ στέρεα ραχοκουκαλιά. Και γι' αυτό λέω ήδη εξ αρχής, εάν η προσφορά δεν είναι επαρκής, το Κοινοβούλιο θα πει τότε ότι θα πούμε όχι. Εγώ είμαι διατεθειμένος να προχωρήσω μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται να καθίσουμε να συζητήσουμε για αριθμούς που είναι κάτω των ανωτάτων ορίων του 2013 διότι αυτά απορρέουν ήδη από τη συνθήκη. Βέβαια τίθεται το θέμα ορισμένων ανακατανομών. Τι θα κάνουμε και με τις ε, νομοθετικές αρχές, διότι δεν μπορεί να μην έχει νομοθετική, ε, νομική βάση μάλλον το, το κάθε κονδύλι. Όμως, όπως μας είπε και η διαπραγματευτική εντολή της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, αυτά βασίζονται όλα στις διατάξεις της συνθήκης. Έτσι λοιπόν πρέπει συζητώντας και με τα Συμβούλια Υπουργών των διαφορών χαρτοφυλακίων δηλαδή, πρέπει να αντιληφθεί και το Συμβουλίο ότι έχει κοινό συμφέρον με το Κοινοβούλιο να μην επιτρέψει τα θέματα αυτά να κρυθούν σε άλλο επίπεδο, αλλά να προχωρήσει σε μια διαδικασία συναπόφασης και όχι μονάχα υπό την πίεση των αριθμών. Έτσι λοιπόν ο κύριος Σέρκας έχει δίκιο ότι είναι εδώ και θέμα θεσμικής αντιπαράθεσης. Η κυρία Μπάουερ μίλησε για το θέμα του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και για την χρήση του στη γεωργία. Όπως και για άλλα θέματα και η Περιφερειακή Επιτροπή και η Επιτροπή ε, μεταφορών συζητούν την διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Έτσι και εσείς πρέπει να συζητήσετε με την Αγροτική Επιτροπή για, το, για την πτυχή αυτή του θέματος. Και αν ίσως προτείνετε κάτι διαφορετικό, ώστε ας πούμε να ληφθεί υπόψη η πτυτικότητα αυτή των τιμών στις παγκόσμιες αγορές, η αστάθεια δηλαδή. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αν πείτε εσείς ότι η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να συμπαραταχθεί μαζί σας για την ΑΒ πτυχή της ε, νομοθετικής διαπραγμάτευσης, τότε εμείς θα είμαστε stand-by. Αλλά από μόνοι μας δεν πρόκειται να αναλάβουμε σχετική πρωτοβουλία, διότι εμείς σεβόμαστε απολύτως τα προνόμια των κοινοβουλευτικών επιτρόπων. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για το MFF, είμαστε αρμόδιοι για την διαθεσμική διαπραγμάτευση και για την διαχείριση ολόκληρου του προπολογισμού, που είναι βέβαια πάρα πολύ τεχνικό πρόβλημα, αλλά και πολιτικό ταυτόχρονα. Και αν εσεί έλθετε και μα πείτε τώρα να σα συνοδεύσουμε στην Α ή Β διαπραγμάτευση, τότε θα το πράξουμε. Αλλά δεν θα αναλάβουμε μόνοι μα εμεί τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Διότι αλλιώ θα φτάσουμε σε μια σύγχυση ε, των θεμάτων που ασφαλώ για αυτήν θα μπορέσει να μα επικρίνει το Συμβούλιο. Για την κυρία Σρέντερ το εργαλείο Progress. Με βρίσκει σύμφωνο η παρατήρησή σας, αλλά και το σύνολο των αριθμών που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Μεγάλος αριθμός κονδυλίων που δεν πρόκειται να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, όπου δηλαδή έχει κάποια προνόμια η Κομισιόν ή το Συμβούλιο να διαχειριστεί κάποια κονδύλια Δηλαδή, ποια θα είναι τα ποσοστά των πιλωτικών προγραμμάτων, ποια θα είναι άλλων μέτρων, σε ποιε κατηγορίε θα υπαχθούν κτλ. Αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευση. Εδώ δεν υπάρχουν ακόμα τα συγκεκριμένα νούμερα. Και επομένω, εφόσον θέλουμε να τα αναλύσουμε αυτά και να τα περιλάβουμε, θα χρειαστεί αυτό να το κάνουμε πλέον στη βάση άλλων λογαριασμών που θα μας υποβάλει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική επιφύλαξη. Εδώ ομολογώ ότι βρίσκομαι σε δυσχερή θέση, διότι αφενός στην Επιτροπή Σούρε είχε υπάρξει κάποια διατύπωση που ήταν κάπως ε, δυσχερής για μας. Αλλά θα σας πω τώρα από το δικό μου Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, όταν πήγαινα, το Bundesrat, το γερμανικό δηλαδή, όταν πήγαινα στην Ελλάδα, ότι δεν ε, είναι δυνατόν να παραβλεφθεί η υπερχρέωση. Και η δική μου, το δικό μου ομοσπονδιακό κρατήδιο έβαλε πρώτο στο Σύνταγμα την ε, απαγόρευση υπερχρέωσης. Συνδέονται οι βοήθειες από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για μας, το Σλέζι Χόλσταϊν δηλαδή, με την απαγόρευση υπερχρέωσή μα, Εφόσον την παραβούμε, κόβονται τα κονδύλια από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Για τη δική μας, για το δικό μα Ομοσπονδιακό Κρατήδιο, το Σφέλεζι Χόλσταϊν. Τώρα βέβαια η προσωπική μου γνώμη είναι εξή. Εάν θέλουμε να πετύχουμε κάποια νούμερα, για να πρέπει να μιλήσουμε για ορισμένες ιδιότητες προγραμμάτων. Δεν μιλώ τώρα ειδικά για την μακροοικονομική επιφύλαξη, αλλά τι θα κάνουμε με τα προγράμματα, πού θα βάλουμε το κέντρο, τα κέντρα βάρους, πού μπορώ να πείσω χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς να χρηματοδοτήσουν κάποια προγράμματα που να μην είναι αυτά που αρέσουν σε κάποιες κυβερνήσεις, αλλά να είναι αυτά τα οποία προσφέρουν κάτι στην απασχόληση. Τότε να δοθεί ένα πράσινο φως δηλαδή για την διαχείριση της κρίσης και να μπορέσει να προβλεφθεί κάποια χρηματοδότηση στην πολιτική συνοχής. Σε αυτό το πλαίσιο θα παίξει κάποιο ρόλο ποιος είναι ο προσανατολισμός των ε, ταμείων αυτών, ποια είναι η προοπτική τους να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Αν το πετύχουμε αυτό νομίζω θα έχουμε επιτύχει σημαντική πρόοδο και θα έχουμε και μια στέρεη θέση και απέναντι στην ε, κοινή γνώμη, η οποία καμιά φορά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ευχαριστώ. Κάλφιν. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ίσως ε, διαφωνώ λίγο όσον αφορά τη μακροοικονομική επιφύλαξη. Αλλά ίσως να μην είναι εδώ κατάλληλος τόπος για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Bon, euh, nous voyons que nous avons une... Βλέπω εδώ ότι έχουμε μια διαπραγματευτική ομάδα αρμονική. Καλό είναι φυσικά να διατυπώνονται οι διαφορές, ε, αλλά βλέπει κανείς καθαρά. Γνωρίζουμε αυτό το είδος άσκησης. Υπάρχει μια θεσμική πτυχή και μια πολιτική πτυχή και οι διαχωριστικές γραμμές ε, υπάρχουν και ίσως οι κατευθύνσεις δεν είναι πάντα ίδιες. Ε, πιστεύω ότι στο πλαίσιο όλων των ανταλλαγών που έχετε και το φόρτο εργασία σα είναι πολύ σημαντική και αυτή η άσκηση διότι εδώ τα μέλη αισθάνονται ότι ε, σχετίζονται με αυτή τη σημαντική διαπραγμάτευση και εσείς μπορείτε να ακούσετε κάποια σχόλια από αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη επιτροπή η οποία έτσι συμμετέχει. Θα το λέμε σε όλες τις επιτροπές. Ε, σας το λένε αυτό πιθανώς σε όλες τις επιτροπές από τις οποίες περνάτε. Όταν βλέπουμε το διακύβευμα της επόμενη. Ε, του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου το κείμενο για το οποίο μιλάμε, δεδομένο των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένων και των προσδοκιών των συμπολιτών μας, ε, πιστεύω ότι εδώ η πρόκληση είναι γιγάντια. Και εμείς ε, βασιζόμαστε στην ικανότητά μας για συμβιβασμούς αλλά και στη δική σας υποστήριξη ώστε να μην έχουμε την νύχτα των μεγάλων μαχαιριών αλλά των μεγάλων αριθμών ώστε όλα αυτά να έχουν ευτυχές αποτέλεσμα και η αποφασιστικότητα που διατυπώνεται σήμερα να εκπληρώσει τους στόχους σας. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Euh, Ωραία λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και δίνω το, δίνω λόγο στην κυρία Μογάν Σαχτιέ ε, επεκτείνοντας έτσι τη συζήτηση που μόλις ε, κάναμε για το σημείο 5 που αφορά το σχέδιο έκθεσης ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω πριν δώσω τον λόγο στην κυρία αυτή ότι θα αντιστρέψουμε δύο θέματα του ημερήσια διάταξη. Ζητώ συγγνώμη και κυρίω τον εισηγητή και τον κύριο Κόζα. Όπω ξέρετε, στι 6 ώρα πρέπει να φύγω για να συζητήσω τον εισηγητή, ε, με τον συνεισηγητή προπολογισμών για τη διαπραγμάτευση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Εφόσον συμφωνεί λοιπόν ο κύριο Κόζα, θα αντιστρέψουμε τα σημεία 6 και 7. Η κυρία Ήξ λοιπόν θα προεδρεύσει τις εργασίες μας στις 6. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κυρία Μωράν ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που σας υποβλήθη η συζήτηση σήμερα προέρχεται απευθείας από τις εργασίες που εμείς πραγματοποιήσαμε στην ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Εγώ προσπάθησα να ενσωματώσω όσο το δυνατόν καλύτερο όσα υπόθηκαν παραμένοντας ανοιχτή σε οποιασδήποτε επιπλέον προτάσεις. Καταρχάς πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσω πως η έκθεση που σας προτείνεται εδώ έχει συνταχθεί υπό το πνεύμα της ενίσχυσης μιας απαραίτητης επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο για τη διατήρηση σε αυτές τις εποχές κρίσης της ευρωπαϊκής δυναμικής, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την προσαρμογή των μισθωτών στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων και για την προετοιμασία τους για την εξέλιξη των θέσεων εργασίας προβλέποντας αυτές τις εξελίξεις. Αυτή η εξέλιξη και αυτές οι προβλέψεις Αυτές οι προσδοκίες ε, δεν είναι άσχετες με τη βούλησή μας, ε, με τη βούληση που έχουμε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να διαθέσουμε στο πιο έθραυστο, στους πιο έθραυστος πολίτες ε, αποτελεσματικές πολιτικές ένταξης αυτών των έθραυστων πληθυσμών ή επανένταξης ενσωματώνοντας ταυτόχρονα το νέο θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας που πλέον εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα σημεία τα οποία θελήσαμε να ε, τονίσουμε περισσότερο σε αυτή την έκθεση. Το πρώτο σημείο, το οποίο για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο, αναπόφευκτο και ουσιώδους σημασίας από πολιτική απόψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να συμμετέχει στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Ευρώπης 2020. Υπό αυτή την νόημα αυτή την πολιτική συνοχή της Ευρώπης 2020 δεν πρέπει να την αναλύσουμε σε τέτοιο βαθμό που να υλοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο χωρίς να υπάρχει αυτό το όραμα του συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε με καλά, πολλοί από σας το γνωρίζετε. Έχουν σημαντικές πιέσεις ε, από αμφότερες τις πλευρές για την περιφερειοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο ένα ή στο άλλο επίπεδο, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι συμφωνούν ε, όλες οι πολιτικές ομάδες ότι αυτή η πολιτική κοινωνική συνοχής εντάσσεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα και συνεπώς αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να προσέξουμε, να διατυπώσουμε πολύ σωστά τις λεπτομέρειες των διαφόρων τροπολογιών μας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο ήθελα να επιμείνω είναι η ε, επιφύλαξη, η ρησιμότητα. Μιλήσαμε για αυτήν, για το, όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η μακρονομική επιφύλαξη, για την οποία έχουμε μιλήσει εκτενώς σε διάφορες πολιτικές ομάδες, αποτελεί πραγματικά κάτι που πρέπει να προωθήσουμε σε κοινωνικό επίπεδο επειδή αποφέρει αποτελέσματα για τους πιο εύθραυστους πληθυσμούς στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Τέλος, ένα σημείο που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές, θέλω να σε επισημάνω την αποτελεσματικότητα με την απαραίτητη με τον ε, την απαραίτητη εκτίμηση επιπτώσεων, την ορατότητα την, το ευανάγνωστο χαρακτήρα ας πούμε αφορά την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει αυτή η δυνατότητα ε, εύληπτης πολιτικής να υπάρχει στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σήμερα παρακολουθώντας ε, την εφαρμογή στο ένα ή στο άλλο κράτος μέλος αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι δεν γίνεται μέγιστη αξιοποίηση και ότι έτσι ορισμένα άλλα ταμεία λειτουργούν με τα χρησιμοποίητα υπόλοιπα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι καταστροφικό και δεν είναι κάτι που επιθυμούμε σε περίοδο κρίσης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλέψουμε πολιτικές ε, ε, αρρωγής προς τους ε, διάφορους παράγοντες ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να διευκολύνουμε τη χρήση, την αξιοποίηση αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πιο γρήγορε πληρωμές, αρρωγή προς τα κράτη-μέλη ώστε οι μερικές πληρωμές να είναι επίσης δυνατές. Αυτό προβλέπεται στο κείμενο. Θα πρέπει να γίνεται και στην πράξη. Και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε απλοποίηση των φακέλων για τα χαμηλότερα ποσά που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βλέπουμε ότι συχνά οι μικροί φάκελοι μικρού πεδίου εφαρμογής. δεν έχω καμία σχέση με το Φεντέρ και το Φεντέρ. Θα πρέπει λοιπόν να απλοποιήσουμε αυτούς τους φακέλους ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ένα από τα σημαντικά σημεία που αναφέρω επίσης και στις ε, και η ένταξη των κοινωνικών εταίρων. Με την ένταξη των κοινωνικών εταίρων στην χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου επιθυμώ να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά και την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ενδεχομένως ε, να του δεσμεύσουμε ένα κομμάτι ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. Άκουσα ε, προλίγου την κυρία Στάιντρουκ η οποία πρότεινε διεθνικές συνεργασίες ε, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών των πολιτικών πιστεύω ότι θα χρειαστεί και αυτό να μας αποσχολήσει όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέλος, προτείνουμε την κεφαλαιοποίηση με οδηγούς βέλτιστων πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί μια κοινωνική πολιτική, ένα σύνολο κοινωνικών πολιτικών για την αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό το λόγο θα πολεμήσω μαζί σας κυρία Πρόεδρε ώστε αυτό το κοινωνικό ταμείο να παραμείνει ξεχωριστό από τις περιφερειακές πολιτικές παρότι πρέπει να συντονίζεται με αυτές και να παραμείνει μια αποτελεσματική πολιτική απασχόληση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Κίνγκα Κούντς ε, πρώτα απ' όλα. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα Χαιρετίζω αυτό το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ. Θεωρώ ότι συνάδει ιδιαίτερα με τον τρόπο σκέψης ε, που όπως εκφράστηκε στην ε, ομάδα εργασίας και αυτό φαίνεται στο κείμενο. Θέλω να αναφέρω κάποια σημεία. Θα το σχέρουμε ιδιαίτερα ε, για το γεγονό ότι ζητάτε να υπάρχει πολιτική προτεραιότητα για το ESF και να διατηρηθεί το 25% μερίδιο κοινωνικής συνοχής ε, στα πλαίσια του ESF, θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το μερίδιο. ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια για αυτούς τους στόχους. Και ακούγοντας, ε, αν θέλετε και όσα διαμήθησαν νωρίτερα, συζήτηση για το MFF, ναι, εσείς μιλάτε για την ε, μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση λόγω της εμπειρίας που έχουμε αντιλήσει από τις δυσκολίες των κρατομερών να προσαρμοστούν ε, στους δημοσιονομικούς κανόνες και λέτε και ότι θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν ε, στην προετοιμασία της νομοθεσίας και στην παρακολούθηση αυτής και να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση κτλ. Ναι, αυτά είναι πολύ σημαντικά και ε, εξίσου σημαντικά στοιχεία, ενδιαφέροντος για όλους όπως ακούστηκε ο σταμάτα Αυτό όμως που θα ήθελα να δω πιο ρητά στο κείμενό σας, είναι το εξή. Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι η άρση όλων των μορφών διακρίσεων είναι σημαντική δικό. Ναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το πούμε πιο ρητά. Να μην δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ από ε, σε προγράμματα που ε, σε έναν βαθμό προωθούν την διακριτική μεταχείριση και τον αποκλεισμό. Γιατί έχουμε τέτοια παραδείγματα στην προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο. Στην ε, ομάδα εργασία συζητήσαμε μακρόν το θέμα του θεματικού συγκεντρωτισμού και κατά πόσον είναι σε καλό επίπεδο, είναι υπερβολικό συγκεντρωτισμό, είναι λίγος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πέρα από το να ορίσουμε τους αριθμούς των στόχων, να ορίσουμε τους στόχους σε αριθμούς, πιο σημαντικό είναι να έχουμε μια γενική εικόνα του σε ποιο βαθμό ο, η επιλογή των θεματικών νοτήτων καλύπτουν γεωγραφικά τα κρατημέλη και όλους τους στόχους, π.χ. στρατηγικές ε, ε, για τους Ρωμά, που αφορά πολλά κράτη-μέλη. Στρατηγικές απασχόλησης παιδείας, θεματικές στρατηγικές λοιπόν που αφορούν κρατημέλη. όλα τα κρατημέλη. Ναι, μεν λοιπόν θεματική συγκέντρωση, αλλά θα πρέπει να συνδυάσουμε τις θεματικές ενότητες με τις εθνικές στρατηγικές. Γιατί ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετά θα πάνε και θα περάσουν σε εθνικές στρατηγικές. Έπειτα, πέρα από τους δίκτες για την απασχόληση και εκπαίδευση, η κοινωνική συμμετοχή και η μείωση της φτώχειας είναι εξίσου στόχοι αυτών των ταμείων. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και τέτοιοι μετρήσιμοι δείκτες της φτώχειας, της κοινωνικής ένταξης, κοινωνικού αποκλεισμού αν θέλετε. Πρέπει να δουλέψουμε και για τέτοιους δείκτες. Επίσης μιλάτε για συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων. Ναι. Για μένα μια πολύ σημαντική ε, συμπληρωματικότητα είναι μεταξύ του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι καλό λοιπόν να φανεί αυτό στο κείμενό σας γενικότερη χρηματικότητα προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από περισσότερα από ένα ταμείο. Μόνο αν υπάρχει συμπληρωματικότητα θα έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των κονδυλίων. Δεν αρκούν βεβαίως ποτέ από όλα τα, τα, τα, τα, κονδύλια, ποτέ δεν είναι αρκετοί οι πόροι, αλλά καλύτερα να τους χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και από τη δική μου πλευρά ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εισηγητρία για την εισηγησή της, για την εκθεσή της που περιλαμβάνει σημαντικά θέματα που έχουμε άλλωστε συζητήσει στην ομάδα εργασία μας. Την ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Συμφωνώ άλλωστε μαζί σας σε ό,τι αφορά αυτή την ορατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η οποία οφείλει να διατηρηθεί έτσι ώστε ειδικά οι πολίτες επιτόπου να γνωρίζουν και ποια είναι τα θετικά τα οποία του έρχονται από τις Βρυξέλλες. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει αυτή, να διατηρηθεί αυτή η ορατότητα του Ταμείου. Τώρα για τα παιδιά που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Όχι μόνο η μείωση αλλά και η πρόληψη. Όχι μόνο η καταστολή αλλά και η πρόληψη είναι πολύ σημαντικά. Καθώς και η διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας. Επίσης ένα θέμα το οποίο πρέπει να περιληφθεί. Συμφωνώ άλλωστε μαζί σας και νομίζω μάλιστα ότι αυτό, αποτελεί και μια ορθή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δηλαδή οι χώρες μέλη οι οποίες διαθέτουν ή οφείλουν να δώσουν χρήματα στα προγράμματα όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή να έρχονται τα χρήματα στις χώρες μέλη. Δεν θέλουμε κάποτε να λάβουν οι απολύπτες τα ε, χρήματα που δικαιούνται, πρέπει να τα έχουν στη διάθεσή τους σύντομα για να μην υπάρχουν κενά. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για μένα είναι σχετικά με, τις, με την χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων. Εδώ προτείνεται το 80% των χρηματοδοτικών κονδυλίων να χωρίζονται το πολύ σε τέσσερις προτεραιότητες στις πιο ε, προχωρημένες περιοχές, περιφέρειες. Αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικός περιορισμός. Εγώ νομίζω πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξουν περισσότερες προτεραιότητες ή από την άλλη μεριά ενδεχομένως ε, διαζευτικά δηλαδή το ποσοστό του 80% να μειωθεί. Για παράδειγμα και σε μεγάλες χώρες όπως τη Γερμανία οι διάφορες περιφέρειες έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες. Άρα να υπάρξει κάποια διαφορετική ε, προσέγγιση. Να υπάρξει μια ευελιξία δηλαδή. Εν τέλει, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Η μακροοικονομική όρη δηλαδή. Και εδώ λοιπόν είμαστε κάπως πιο εύκαμπτοι. Όχι αυτοί που υφίστανται τα μεγαλύτερα δεινά να τιμωρούνται και από πάνω. Αν όμως οι χώρες μέλη πραγματικά αρνούνται να κάνουν κάποια προσπάθεια, κάποια πρόοδο στο θέμα της υπερχρέωσης. Τότε βέβαια θα πρέπει να σκεφτούμε αν ίσως αυτή είναι και η τελευταία λύση, η τελευταία μας δυνατότητα, δηλαδή να προχωρήσουμε σε κάποιες περικοπές. Όχι με την αιτιολογία ότι μια χώρα είναι υπερχρεωμένη. Αν δούμε ότι οι κυβερνήσεις δείχνουν μια θέληση, τότε για μένα δεν είναι θέμα. Αν όμως δούμε ότι μια κυβέρνηση πραγματικά αγνοεί οτιδήποτε της λένε, δεν προχωρεί σε καμία προσπάθεια, τότε ίσως αυτό είναι ένα μέσον για να ασκήσουμε και κάποια πίεση έτσι ώστε να ανταποκριθούν και στις απαιτήσει που τους επιβάλλουν οι Βρυξέλλες. Η ε, κυρία Σρέντερ. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ ιδιαίτερα την εισηγήτρια για την έκθεσή της, η οποία περιλαμβάνει και πολλές από τις προτάσεις που υποβάλαμε και εμείς. Και εδώ τονίζω και πάλι ότι συνεργάστηκε η συγκίτρια με θαυμάσιο τρόπο μαζί μας και πραγματικά εγώ χαίρομαι που θα συνεργαστώ, θα συνεχίσω τη συνεργασία αυτή μαζί της. Τώρα έχω τρία πράγματα. Πρώτο, αυτό που είπε η κυρία Χίρς και που εννοούσα εγώ όταν ρώτησα προηγουμένως τον Επίτροπο σχετικά με τα ποσοστά αν θέλουμε να έχουμε μία δυνατότητα αυτά τα 25% να τα περάσουμε με το 25 ή 50%. Αν θέλουμε δηλαδή να εμείνουμε σε αυτό το 25% για ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, πρέπει μέσα στον κανονισμό του EFSF να έχουμε περισσότερες δυνατότητες να επιτύχουμε κάποιες συμμαχίες. Δηλαδή τότε αυτοί που θέλουν περισσότερα χρήματα του ESF και θέλουν να τα περάσουν τα κονδύλια αυτά, χρειαζόμαστε να έχουμε μια ευκαμψία για να πετύχουμε αυτές τις συμμαχίες. Τότε στο άρθρο 4.3 δεν εξυπηρετούμε το σκοπό μας και διαρθρωτικά είναι λάθος το άρθρο αυτό 4.3. Αν τα εξετάσουμε αυτά σε σύγκριση με τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία θα δείτε ότι εκεί είναι διαφορετικές οι προσεγγίσεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το άρθρο αυτό 4.3, όπως είπε και η κυρία Χίρς, δεν επιτρέπεται να παραμείνει στο επίπεδο της προτεραιότητας των επενδύσεων. Πρέπει να έρθει στο επίπεδο των θεματικών, όπως και ο ΕΦΡΕ, δηλαδή να βάλει αυτές τις 11 προτεραιότητες του γενικού κανονισμού που έχουν τις ε, επικεφαλίδες α, β, γ, δ κλπ. Και για μας είναι οι προτεραιότητες 8, 9, 10. Εκεί πρέπει να γίνει η συγκέντρωση. Αυτό θα σημαίνει ότι στους τομείς εκείνους όπου Υπάρχει ανάγκη στι διαφορέ χώρε μέλη. Να πούμε, ο τομέας 8 απασχόληση, ο τομέα 9 κοινωνική συμπερίληψη κατά πολέμηση φτώχεια και ο τομέας 10 εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Για αυτά τα τρία πρέπει να πάνε τα 80% που σημαίνει συνολικά 16 προτεραιότητες επενδύσεων. Και το υπόλοιπο θα αποτελέσει αυτό το περιθώριο που για τις χώρες εκείνες μέλη που θέλουν να βάλουν αυτές τις κατά μέσον όρο προτεραιότητες το άρθρο 3 και πρέπει να εξελίξουν τις ε, διοικήσεις τους, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε ορισμένες χώρες μέλη, εκεί θα έχουν δυστυχώ το 60%. Εγώ θα ήθελα να βάλουμε εδώ ένα at least. Είναι δυνατόν δηλαδή μια χώρα μέλος να θέλει να διαθέσει το 95% σε αυτές τις τρεις προτεραιότητες που είναι σημαντικά δηλαδή για την κοινωνική απασχόληση για την κοινωνική πολιτική συγγνώμη και για την απασχόληση. Αυτά. Άλλωστε νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη πολιτική αυτή που θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μέσω του ESF. Δεύτερο θέμα. Το άρθρο 6. Χρηματοδότηση των συνεργασιών. Εγώ έχω εξετάσει το θέμα γιατί συντάσσω και κάποιες τροπολογίες. Το πρόβλημα μεγάλο αυτό του άρθρου πρώτου δηλαδή. Γιατί αυτό που απαιτούμε από τους εταίρους είναι να πάνε σε κάθε διοίκηση η οποία διαθέτει χρήματα των διαφορετικών ταμείων να ζητιανέψουν κάποια χρήματα για να φτιάξουν μια δομή για να μπορέσουν να έρθουν στο επίπεδο και να συνομιλούν δηλαδή σε ίδιο ίσο επίπεδο με τις διοικήσεις. Για κάθε λοιπόν προτεραιότητα θα πρέπει να πάνε να ζητιανέψουν χρήματα. Εγώ είμαι αντίθετη. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη διαδικασία η οποία θα, την οποία θα διχειρίζεται μια κεντρική αρχή. Αλλιώ δεν πρόκειται να γίνει καμία συνεργασία, δεν πρόκειται να γίνει καμία εταιρική σχέση. Δεν θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή η δυνατότητα και θα υπάρχουν και χιλιάδε προκαταλήψει που θα προβάλλει κάθε διοικητική αρχή για να μην του δώσει τα λεφτά. Άρα εδώ χρειάζεται κάποια αλλαγή. Η δυσκολία προκαλείται εδώ από τον γενικό κανονισμό που συνδέει τις προτεραιότητες με τους άξονες αυτούς και είναι ένα βασικό πρόβλημα νομίζω μέσα σε όλο αυτό τον τομέα των διαθωτικών ταμείων που εγώ το επεξεργάζομαι γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Το τρίτο είναι το άρθρο 12 για τις λεγόμενες ITI που είναι το εργαλείο εκείνο που επιτρέπει μία ολοκληρωμένη πολιτική στα αστικά κέντρα. πολέμηση της στόχιας και ταυτόχρονα επενδύσεις του ΕΦΡΕ, δηλαδή μικρές αστικές επιχειρήσεις, η υποδομή της πόλης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δηλαδή διασυνδέονται στην περίπτωση αυτή. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένα 5% να πάει κατευθείαν στους Δήμους για να μπορούν να εγκρίνουν αυτοί έργα. Αυτό έχει κάποιο νόημα, διότι ένα τέτοιο αστικό κέντρο μπορεί καλύτερα να επιλέγει μόνο του τα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσει και όχι να γίνεται στο εθνικό επίπεδο. Για το ΕΦΡΕ προβλέπεται, για το ESF προβλέπεται αλλά χωρίς ποσοστό. Μπορεί δηλαδή να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου η συγκεκριμένη πόλη να μπορεί να εγκρίνει για το ΕΦΡΕ κονδύλια, αλλά για το ESF που να πρέπει να πηγαίνει να ζητάει από την εθνική διοίκηση. Γι' αυτό λέω εγώ τουλάχιστον 5%, έτσι ώστε οι πόλει, οι δήμοι δηλαδή, να μπορούν να δαπανίσουν τα χρήματα και από τα δύο αυτά ταμεία. Αυτά. Ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να σα ασκήσω πίεση, αλλά ήθελα να προσθέσω τη θέση μου για τι τροπολογίε, για το κοινοψήφισμα πριν σα αφήσω και αφήσω την Προεδρία στην κυρία Χέρι. Κυρία συγγήτρια στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού ήθελε επίση να μιλήσει και μετά κύριε συγγήτρια, μπορείτε να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Ήθελα να επιμείνω σε δύο στοιχεία αυτού του κανονισμού η εγκατάλειψη του σχολείου είναι μεγάλο ένα πρόβλημα και χαιρόμαστε που συμπεριλαμβάνεται και η σημασία της καταπολέμησης της ενεργειάς των νέων. Έχω κάποιες επιφυλάξεις. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι στον τρέχοντα κανονισμό 2007-2013 αναφερόταν το πρόγραμμα EQUAL που αφορά την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της διακρίσεων στον χώρο εργασίας και που δεν εμφανίζεται στη νέα πρόταση, το οποίο θεωρώ είναι κρίμα. Τέλος, όσον αφορά τον πολιτισμό, δεν παρουσιάζεται ως στόχος κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, θεωρώ ότι συμβάλλει με πολλούς τρόπους στην εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης τεχνογνωσίας και ικανοτήτων και στην οικονομική ανάπτυξη μέσω των βιομηχανιών του πολιτισμού καθώς και στην ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων. Όλο αυτό δεν αναγνωρίζεται επαρκώς και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ρήτα ότι θα πρέπει τα πολιτισμικά στοιχεία να βρουν τη θέση τους ε, σε αυτό το μηχανισμό, ε, για παράδειγμα στο άρθρο 3. Ε, η κυρία Συγήτρια, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, και όλες τις συναδέλφους ε, που συμμετείχαν στην ομάδα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και που ήρθαν επιμελώς εδώ και πολλούς μήνες για να συνεργαστούμε σε αυτό το ζήτημα ώστε όλοι μαζί να καταλήξουμε σε αυτό το νέο κείμενο τη νέα πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτό εξηγεί το πώς εδώ μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά με μια ίδια φωνή όλες μαζί για αυτό το ζήτημα. Σημείωσα όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν, ε, ειδικότερα όσον αφορά το 25% για τις πολιτικές συνοχής, όπως είπε η κυρία Γκέντσκ, το γεγονός ότι πρέπει να αποφύγουμε με ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την ενίσχυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Συνεπώς ε, να εστιάζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε εθνικό επίπεδο σε σημαντικές θεματικές πολιτικές όπως η Ρωμά, η παιδεία και το καθεξής. Όλοι συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν δείκτες μείωσης της φτώχειας και ότι είναι απαραίτητη συμπληρωματικότητα των ταμείων εφόσον αν συντονίζονται σωστά και συνδυάζονται σωστά και δεν παρεκκλίνουν προς και, και εφόσον εφαρμόζονται σε κοινωνικές εφαρμογές. Σημειώσα όσο είπε η κυρία για την πρόληψη της ε, ε, εγκατάλειψης του σχολείου χωρίς κάποια ειδίκευση όσον αφορά την αυστήρη πλευρά της θεματικής συγκέντρωσης ώστε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάποια ε, ευελιξία και όσον αφορά την επιφύλαξη της δυνατιαχής είμαι βέβαιη ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα μπορεί ενίοτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να είναι αιτιολογημένη Εμεί υποστηρίζουμε εξαιρετικά κοινωνικέ θέσεις. Πιστεύουμε ωστόσο ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε δύο φορές ε, τους ε, πιο φτωχού που δυσκολεύονται να ενταχθούν ε, επαγγελματικά. Σημειώσα όσα είπε η κυρία Σρέντερ για το 25% για την πολιτική συνοχής όσον αφορά τις συνεργασίες επίσης και όσον αφορά και τις θεματικές συγκεντρώσεις. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω δεδομένου του έργου που έχουμε ήδη κάνει όλοι μαζί για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τρόπο συλλογικό. Προτείνω μία από κοινού συνεδρίαση όλων των σχεδόν εισηγητών ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το ίδιο πνεύμα και να βελτιώσουμε όλοι μαζί ό,τι μπορούμε να βελτιώσουμε μαζί και μετά ο καθένας από την πλευρά του θα πράξη ανάλογα με τις πεπιθήσεις του. Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεση όλων για τη συνέχιση της εργασίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι πρέπει να διατηρήσετε την ε, ε, κινητικότητα αυτή με την ίδια αποφασιστικότητα όπως και για την εκθέση του κυρίου Κόζα που θα καθορίσει την πορεία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αλλά είμαι βέβαιη ότι ήδη το έχετε αυτό στο νου σα. 16 Μαΐου, 12 η ώρα το μεσημέρι, η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα τις εξετάσουμε 20 και 21 Ιουνίου με συζήτηση για τις τροπολογίες συμβιβαστικέ 10 Ιουλίου και ψηφοφορία στις 10 Ιουλίου επίσης για έγκριση στην Ολομήλεια του Σεπτεμβρίου. Περνώντα το σημείο 7 της σα διάταξης, όπως συμφωνήσαμε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη θέση μου για τις διάφορες τροπολογίες πριν δώσω το λόγο, πριν δώσω τη, συγγνώμη, την Προεδρία στην αντιαχείριση. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοβουλία που είχαμε αναλαβεί εμείς ε, ως συντονιστές ε, για την ε, επαναδρομολόγηση δεδομένου του παλαιότερου έργου της Επιτροπής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρίως με την εκθέση της κυρίας Τούρινεν και όχι μόνο για το ζήτημα των ευκαιριών που προσφέρονται στους νέους σήμερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαμε επιθυμήσει να απαντήσουμε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης του περασμένου Φεβρουαρίου ενσωματώνοντας τα στοιχεία της ακρόασης που έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο στην Επιτροπή μας. Όσον αφορά αυτό το ζήτημα υπάρχουν τρεις προτάσεις ε, τροπολογιών που δεν σας προτείνω να ε, εγκρίνετε. Θα δούμε τι θα ψηφιστεί αύριο στη Δανία. Ωστόσο, κατά την απόψή μου, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα υπέρα. Έχουμε και μια σειρά τροπολογιών που θέτουν κάποιο πρόβλημα διότι παραποιούν εν μέρη το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Κοιτώντα ε, το περιεχόμενο της ε, πρότασης ε, ψηφίσματος που σας έχει υποβληθεί το κυρίως μήνυμα βασίζεται στην ιδέα δημιουργίας μιας εγγύησης για τους νέους βάσει πραγμάτων που υπάρχουν ήδη σε κάποια κρατημέλη. Αυτή πιστεύω ότι είναι η προστιθέμενη αξία που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό το ψήφισμα, διότι για τους νέους μιλάμε διαρκώς όλη την ημέρα και για τα προβλήματα της ανεργία και κάνουμε ότι κάνουμε κάτι. Αλλά σε ορισμένες υπάρχουν χώρε όπως η Αυστρία όπου υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιτυχής που έχουν υλοποιηθεί εγώ προτείνω ενώ σε άλλες χώρες και όπως το Λουξεμβούργο ε, ετοιμάζονται να ακολουθήσουν αυτό το αυστριακό παράδειγμα μπορούμε βάσει της λογικής του benchmarking να δημιουργήσουμε μία πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο σκοπός μέρη του ψηφίσματος και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών για τη βελτίωση του ψηφίσματος που δεν αποτελούν πρόβλημα για μένα, αλλά για άλλη μια φορά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που κάπως ε, με δυσκολεύουν. Αυτό που έχω να σας προτείνω είναι να σας πω που θα ήθελα να προτείνω συμπληρώσεις ή αλλαγές ε, όσον αφορά την ε, τροπολογία 4 την κυρία Λαμπέρ ε, θα μπορούσαμε να το προσθέσουμε θα μπορούσαμε δηλαδή να συγχωνεύσουμε ε, τις τροπολογίες όσον αφορά την τροπολογία 14 της κυρίας Χίρς αφορά ένα σημείο όπου έχουμε τροπολογία του κυρίου Όρη το, η οποία πηγαίνει πιο πέρα από την τροπολογία της κυρίας Χίρς προτείνω λοιπόν να λάβουμε υπόψη ε, την τροπολογία της κυρίας Χρήσης ως συμβιβαστική τροπολογία, την τροπολογία 14, αντί να δεχθούμε την τροπολογία 13 του κυρίου Ορή. Δηλαδή για το εκτιμώντα ε να θεωρήσουμε ότι η τροπολογία 14 αποτελεί συμβιβαστική, πρωτοβουλία μεταξύ, ε, συμβιβαστική τροπολογία μεταξύ των διαφόρων προτάσεων. Όσον αφορά την τροπολογία 23 τη κυρία Λάμπερ ξανά, η οποία δεν βρίσκεται εδώ, αλλά πιστεύω ότι η κυρία Τύρινεν ή η σρεντερ θα μπορούσαν ενδεχομένω να τη αναφέρουν την πρότασή μου. Η κυρία Λαμπέρ μιλάει για inclusive green και John job bridge growth, εγώ προτιμώ στο τέλος δηλαδή της πρότασης να μιλήσουμε για sustainable και job bridge growth, διότι αυτό καλύπτει το πράσινο ζήτημα, το greening, αλλά συμμορφώνεται καλύτερα με τη βασική μας σκέψη όσον αφορά τις επενδύσεις και την οικονομική πολιτική που θα λάβουν χώρα στο μέλλον. Όσον αφορά την τροπολογία 28, για να ευχαριστήσω τον κύριο Όρη ο οποίος όμως έχει φύγει. Ε, θα προτείνω ξεχωριστή ψηφοφορία αποδεχόμενη το πρώτο κομμάτι της τροπολογίας του και απορρίπτοντας το δεύτερο κομμάτι, διότι στο δεύτερο διαγράφει την αναφορά στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις που εγώ δεν μπορώ να δεχτώ εύκολα. Όσον αφορά την τροπολογία 31, σας προτείνω και εκεί μία τροπολογία με ξεχωριστή ψηφοφορία για να ευχαριστήσω τον κύριο Καμπρινόχ. Εάν θέλετε να το δεχθείτε, το πρώτο τμήμα, το πρώτο κομμάτι δηλαδή θα είναι is convinced. Εδώ θα έχουμε δηλαδή μια προφορική τροπολογία και ξεχωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο κομμάτι ξεκινά το is convinced that one effective way of bringing young people back to work consists in introducing in developing systemic reforms in order to tackle structural unemployment. Αυτό θα είναι το πρώτο κομμάτι και εγώ θα είμαι υπέρ αυτού του τμήματο, αντιθέτω, δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσουμε το Introducing More Flexible Labor Laws in the EU National Level. Αυτά είχα να πω για την τροπολογία 31. Και τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 52 και εκεί έχω να σας προ... Α, συγγνώμη, ξέχασα την τροπολογία 41. Για την τροπολογία 41 της κυρίας Χίρς ε, θέλει να κάνει έκκληση στα κράτη-μέλη, ενώ εγώ πρότεινα να κάνουμε έκκληση στην Κομισιόν. Ε, θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε προσθήκη την τροπολογία της κυρίας Χίρς, δηλαδή να κάνουμε έκκληση και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη Συμφωνεί η συντακτρία της ε, τροπολογίας, μπορούμε λοιπόν να το θεωρήσουμε ως προσθήκη, την τροπολογία 41. Και τέλος, ε, όσον αφορά... Α, συγγνώμη, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ακόμα δύο τροπολογίες. Τροπολογία 49. Το ίδιο πρόβλημα πρόκειται για τροπολογία της κυρίας Λάμπερ που ε, παραπέμπει στο Green Economy εγώ θα το άλλαζα με sustainable economy, το green economy στο τέλος της πρότασης. Ε, η τροπολογία αυτή πλησιάζει πολύ στις ανησυχίες του κυρίου Κραπνόχ στην τροπολογία 21. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προσαρμόσουμε τη σύνταξη. Θα το κρίνετε εσείς. Όσον αφορά την τροπολογία 52 του κυρίου Όρη, θα μπορούσα να τη δεχθώ εάν αυτός δεχθεί να υποβάλει μια προφορική τροπολογία που θα επαναλαμβάνει τη δική μου αρχική ε, διατύπωση undermine. Συνεπώς το πρώτο κομμάτι της ε, τροπολογίας 52 θα ήταν calls on the Commission to make sure that all plans and recommendations to member states to regain fiscal sustainability do not destroy or undermine. Δεν καταστρέφουν ούτε υπονομεύουν τις πολιτικές και τα προγράμματα. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Ζητώ ε, συγγνώμη για αυτό το τηλεγραφικό τρόπο ομιλίας μου. Ωστόσο έχουμε τους χρονικούς περιορισμούς ε, με τους οποίους εργαστήκαμε και αφήνω τώρα την κυρία Χίρς να κρίνει το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Ε, σας εύχομαι καλή δουλειά και ζητώ συγγνώμη και τον κύριο Κόζα που δεν θα είμαι παρούσα στην παρουσίαση της έκθεσης του. Ευχαριστώ. Mrs. Turunen. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ. Λίγα σχόλια να κάνω για τις ε, τροπολογίες των πρασίνων. Μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή του όρου green με τον όρο sustainable. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποιες τροπολογίες που θεωρώ είναι συγχυτικές. Πολλές άλλες είναι εξαιρετικές, το λέω. Αλλά υπάρχουν και κάποιες τις οποίες ε, θα αμφισβητούσα. Τροπολογία 11 των συντηρητικών μεταρρυθμιστών λέει ότι οι βασικοί λόγοι της ε, αμερικής των νόμων είναι η συνεχής εξάρτηση από το σύστημα πρόνοιας και από θέματα νοοτροπίας. Ρωτώ, είναι αυτή η κύριοι λόγοι? Ναι, μεν, μπορεί να υπάρχει μια κάποια ακαμψία στην αλλά είναι ο βασικός λόγος και έπειτα η χώρα με το υψηλότερο επίπεδο παροχών κοινωνικών υπηρεσιών σε σχέση με το ΑΕΠ, που είναι η Δανία και οι κατοχώρες έχουν χαμηλό επίπεδο ανεργίας μεταξύ των άνω. Οπότε είναι απλά εσφαλμένη αυτή η διαπίστωση και δεν θα πρέπει να συγκληθεί αυτή η τροπολογία. Τροπολογίες 16 και 17 ε, των φιλελευθέρων και των ρυθμιστών ότι λέει ότι οι νέοι δεν είναι υπεύθυνοι για την κρίση. Ναι, ναι, ναι, δεν το καταλαβαίνω όμως. Οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι δηλαδή, ή μάλλον η, τροπολογία λέει ότι υπάρχει, υπάρχει ε, υπευθυνότητα των νέων, όμως εγώ θεωρώ ότι εφόσον δεν ήταν στην ενεργή αγορά εργασίας και δεν είχαν λάβει ε, ε, κρίσιμες αποφάσεις, πώς μπορούν να είναι υπεύθυνοι. Να διαγραφεί λοιπόν. Έπειτα, πάμε στην τροπολογία 28. Η κυρία Πέρες είπε ότι θα μπορούσαμε να προβούμε σε χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα μάλλον, γιατί υπάρχει θέμα τη συλλογική διαπραγμάτευση, το οποίο θέλει να το κρατήσει η κυρία Πέρε και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Όμω το ΕΛΚ θέλει να διαγραφεί το γεγονό ότι η προσωρινή απασχόληση επηρεάζουν ιδιαίτερα αρνητικά του νέου. Ναι, ρωτήστε τον ΩΣΑ. Ε, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για την υψηλή ενέργεια μεταξύ των νέων. Θα, θα σας πούνε ότι είναι η έλλειψη εμπειρία για την ενισερχόμενη στην εργασία, αλλά και δεύτερον γιατί είναι ε, σε επισφαλείς εργασίες και σε εποχές κρίσης οι προσωρινά απασχολούμενοι είναι αυτοί που είναι σε επισφαλή θέση και χάνουν ε, την αγορά, τη θέση τους μόνο στην οργανωσία. Ζητώ συγγνώμη αν θα προσπαθήσω να επιταχύνω τροπολογία 43. Το ΕΛΚ θέλει να διαγραφεί η δυνατότητα να υπάρχει χωριστός και ειδικό τίτλος για την νεολαία. Ρωτώ, γιατί. Αυτό είναι ένα κομμάτι των συζητήσεων. Και αν κατάλαβα καλά, ίσως να υπάρχει συνένεση από αυτού. Ίσως να ασφάλω εγώ. Αναφέρομαι ε, για το νέο MFF και ένα σχετικό τίτλο για την νεότητα. Και πάλι τώρα, τροπολογία 4 και πάλι το ΕΛΚ. Να μην γίνει αναφορά και στις οργανώσεις των νέων μεταξύ των οργανώσεων ε, που πρέπει να συμπεριληφθούν. Μα γιατί, γιατί να μην γίνει αυτή η συμπεριληψή. Και τέλος τροπολογία 51 όπου θέλει θέλουν να αντικατασταθεί ο όρο decent and quality jobs με τον όρο new jobs. Δεν θέλουμε μόνο νέες εργασίες, αλλά και αξιοπρεπείς ποιοτικέ εργασίες. Δηλαδή θέλουμε ανθρώπου που να μπορούν να βγάζουν τα προστοζήν και να εργάζονται σε καλέ συνθήκε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνει αυτή η διατύπωση. Και ούτω ή άλλως είναι μία γλώσσα που έχει εγκρίνει και η Επιτροπή. More and better jobs, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε είναι κάτι που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε παρότι ζούμε εποχή κρίσης. Πέρα από αυτά λοιπόν τα αρνητικά στοιχεία, πιστεύω ότι κατά τα λοιπά έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Ελπίζω κάποιος εκπρόσωπος του ΕΛΚ κατά κύριο λόγο να μου απαντήσει ή και κάποιος από την ε, ομάδα των ε, συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ähm, Ευχαριστώ. Αύριο μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Και αφού θα ψηφίσουμε αύριο μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως που είναι το υπαριθμό 6. Ας αναλάβει τώρα την διεύθυνση συζητήσεως, ο... μάλλον ας, ας το λόγο τώρα ο κ. Κώσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας συγχαίρω πρώτα και σας ευχαριστώ που είστε παρούσα. Ακόμα μια, σε μια ώρα που είναι σχετικά προχωρημένη. Πάντως είναι χρήσιμο να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων. για αυτή το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει και σχέδιο εκθέσεως, διότι είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι η Επιτροπή μας, απασχολήσεως δηλαδή, αποδίδει μεγάλη προσοχή στο θέμα αυτό. Το μεγάλο ενδιαφέρον που προσήλκησε η έκθεση αποδεικνύεται και από το μεγάλο αριθμό, 89 το σύνολο, των ε, τροπολογιών. Εμείς εργαζόμαστε ήδη εδώ και ένα δίμηνο για το θέμα αυτό και συνεργάστηκα με πολλούς συνομιλητές οι οποίοι με βοήθησαν σε αυτή την προπαρασκευαστική εργασία και του οποίους επιθυμώ να ευχαριστήσω για την ε, συνεργασία τους. Προσπαθήσαμε να εναρμονίσουμε τα διάφορα σχέδια εκθέσεων που συνδέονται στενά με το θέμα. Θα ήθελα να σας δώσω μια επισκόπηση αυτών των 89 τροπολογιών. Ποια ήταν η βάση των ε, τροπολογιών αυτών. Δεν μπορώ βέβαια, δεν θα μπορέσω βέβαια να επισέλθω σε λεπτομέρειες διότι τότε θα χρειαστώ πολύ περισσότερο χρόνο για να το πράξω αλλά θέλω να τονίσω πέντε επιμέρους ε, σημεία. Πρώτον, οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου αυτή η νέα νομοθετική διαδικασία ενισχύει υπερβολικά τον ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν δηλαδή, και εδώ πρέπει να εξευρεθεί κάποια ισορροπία για τις αρμοδιότητες αυτές. Δεύτερο, οι δεσμεύσει των χωρών μελών. Εδώ νομίζω θα ακολουθήσουν ακόμα πολλές συζητήσεις και αρκετές αντιπαραθέσεις. Τρίτο, θέμα της διαδικασίας. Εδώ επίσης νομίζω θα ακολουθήσουν πολλές συζητήσεις, διότι πιστεύω ότι το νομοθετικό κείμενο προβλέπει ως έχει τώρα υπερβολικά πολλές αρμοδιότητες ε, υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτο, επίσης Η ασφάλεια δικαίου. Πολλές άλλωστε τροπολογίες συνδέονται με το θέμα αυτό. Τέλος, ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά ιδιαίτερα λόγω της καταστάσεώς μου, δηλαδή η κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρίες. Νομίζω ότι το σχέδιο αυτό στο οποίο εγκύπτουμε τώρα έχει μεγάλη σημασία για την ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. που έχει ως στόχο να επιτρέψει την πρόοδο των χωρών μελών και αυτή να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Πρόκειται για ένα εργαλείο βάσης και γι' αυτό το σχέδιο που θα υποβάλουμε, το νομοθετικό σχέδιο που θα υποβάλουμε πρέπει να είναι πολύ ισορροπημένο. Δέχομαι ότι στο μέλλον θα είναι απαραίτητο να ενισχυθούν ορισμένοι κανόνες και αναγνωρίζω ταυτόχρονα, έστω και αν αυτό δεν προκύπτει, δεν απορρέει από το νομοθετικό αυτό σχέδιο, Κάθε ένα από τους φορείς που εμπλέκονται έχει τα δικαιώματά του και τις υποχρώσεις του. σε ό,τι αφορά τις υποχρώσει και τα δικαιώματα των χωρών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχει ισότητα και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να επανεξισορροπηθούν οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, τα δικαιώματα, οι των δύο επιπέδων και άλλωστε των χωρών μελών όταν αυτές ποιούνται χρήση των διαφόρων πόρων. Οι διοικητικέ επιβαρύνσεις δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρές. Έχουμε συζητήσει στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου για την διοικητική επιβάρυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει προσπάθεια να μειωθεί αυτή η επιβάρυνση. Από την άλλη μεριά, το νομοθετικό σχέδιο δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλά σχέδια γνωμοδοτήσεων τα οποία στοχεύουν στην γραφειοκρατική ελάφρυνση. Μένει όμως ακόμα δουλειά να γίνει, διότι αυτές οι προαναφερθήσεις 89 τροπολογίες δίνουν κάποιους βασικούς προσανατολισμούς. Τώρα υποθέτω ότι οι συνάδελφοί μου ευρωβουλευτές θα είναι σύμφωνοι ότι θα πρέπει να προσθεθούν και άλλες για να συμπληρωθεί το σχέδιο αυτογνωμοδοτήσεως που απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή αφού θέλουμε να δείξουμε ποιες είναι οι προθέσεις μας. Εν τέλει αναμένω τα σχόλια και τις τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να τοποθετηθούν οι σκιώδεις συγητές και οι συγγήτριε. Πρώτα ο κ. Κουτιέρες Μπριέτο, μετά κ. κυρία Σρέτερ και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κώσα για αυτή την ε, γνωμοδότηση με την οποία ουσιαστικά συμφωνούμε ιδίω γιατί δεν ζητούμε κάτι τόσο απλό και αμεληταίο. Μιλάμε για την καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν άμεσα την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δεν είναι τυχαίο όταν βλέπουμε στοιχεία του Ευρωπαρόμετρου, βλέπουμε ότι συμπίπτουν δύο θεμελιώδη ζητήματα για να κάνουμε εισαγωγή συζήτηση. Αναφέρομαι στι περιφέρειε εκείνες που έχουν λάβει τα πιο πολλά κονδύλια ε, από το Ταμείο Κοινωνική Συνοχή. Είναι περιφέρειε που αγαπούν περισσότερο την Ευρώπη. Είναι πιο φιλευρωπαϊκές περιφέρειες. Άρα λοιπόν η οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών με την πολιτική συνοχή, με την πολιτική απασχόληση που δημιούργησαν εκατομμύρια ε, θέσεων εργασίας και δημιούργησαν πάνω από 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, α, είναι η αιτία που δημιούργησαν αυτό το ρομαντικό συνέστημα του φιλευρωπαϊσμού. Αν μου επιτρέπετε να πατήσω και εγώ στο ερώτημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αγγίζουν ακριβώς το ίδιο το θέμα της ύπαρξης αυτού αυτό το Ταμείο Συνοχής, αναφέρομαι σε αυτό που συζητούμε συνεχώς όλο αυτό το απόγευμα, την μακροοικονομική πολλαπλή συμμόρφωση, την ερεσιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα κονδύλια συνεχίζουν να πηγαίνουν για το σκοπό της αλληλεγγύης, ώστε οι περιφέρειες που υπολείπονται να μπορέσουν μια μέρα να φτάσουν ε, αυτούς που είναι μπροστά. Πιστεύω ότι θα είναι τεράστιο σφάλμα να μετατρέψουμε τη φιλοσοφία του ΣΥΠΑΚ σε κάτι που θα διέπει τα ταμεία της συνοχής. Όχι. Κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μοιράσει μηνύματα στα Αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να σεβόμεθα την πολιτική που ακολουθήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες στα ταμεία συνοχής που διέπονται την αρχή της αλληλεγγύης. Κατανοώ ότι υπάρχουν στόχοι στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ουσιαστικά να τιμωρηθούν περιφέρειες που υπολείπονται στα αριθμητικά στοιχεία. Γιατί αυτοί που τιμωρούνται είναι οι πολίτε, γιατί οι πολίτε είναι που λαμβάνουν τα κονδύλια από το Ταμείο συνοχή, όχι οι κυβερνήσεις που δεν εκπληρούν τους όρους, αν θέλετε, και τι προποθέσει που θα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη η διαφωνία μου. Κλείνοντα, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κώσα σε ό,τι αφορά την απλούστευση. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο προσωπικότητες. Άλλοι είναι αυτοί που συντάσσουν την θεολογική σκέψη μια πρόταση και άλλοι αυτοί που συντάσσουν το διατακτικό με τα άρθρα. Λέει η Κομισιόν ότι ένας βασικούς στόχος είναι η απλούστευση των πολιτικών συνοχής και εγώ την εντύπωση με την πρόταση που βλέπουμε είναι να επιτυγχάνουν το αντίθετο. Αύξηση της ερεσιμότητας, εμείς είπαμε ότι είμαστε κατά της ε, ε μακροοικονομικής ε, και με αυτή την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αιρεσιμότητα απλά αυξάνουμε την γραφειοκρατία, δημιουργούμε μια κατάσταση αδύνατο να είναι αποτελεσματική. Και από πλευράς που να πω ότι αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής. Στα πλαίσια της κοινή στρατηγικής μας η καρδιά πάντοτε ήταν η δημιουργία προσδόντων εργασία. Ναι, μεν αγώνα κατά τη φτώχεια, αλλά κατά κύριο λόγο περισσότερη απασχόληση. Λέει λοιπόν μια πρόταση ότι τα διάφορα κρατημέλη και περιφέρειες μέσα σε ένα κατάλογο 11 στόχων να επιλέξουν και να θέσουν προτεραιότητες μεταξύ αυτών των στόχων με κάποια κριτήρια. Οι περιφέρειες, τα κράτη-μέλη που έχουν ανεργία πάνω από 10% θα πρέπει να θέσουν υποχρεωτικά ως πρώτο στόχο τη δημιουργία απασχόληση, λέω εγώ, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, αυτό θα πρέπει να είναι ο πρώτο και υποχρεωτικό στόχο. Για να περάσουμε ένα καλό μήνυμα. Ότι το μήνυμα το πρώτο δεν είναι δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά δημιουργία θέσεων εργασίας και ή δυνατόν ποιοτικής εργασίας. Αυτά ευχαριστώ. Danke, Elisabeth ähm, κυρία Σρέντερ, εγώ εξέτασα προσεκτικά το σχέδιο του κυρίου Κώσα και βρίσκω ότι προσθέτει κάτι σημαντικό στο σχέδιο της Κομισιόν. Την προσβασιμότητα, ας πούμε, την accessibility για πρόσωπα με αναπηρίες, κάτι για το οποίο είχαμε αγωνιστεί και αυτό βρίσκω ότι το προσθέτει πολύ καλά. Βέβαια, η ιδέα του να φύγουν οι περιφέρειες, αντί φτωχές περιφέρειες να λέει μόνο φτωχοί άνθρωποι, εγώ δεν συμφωνώ. Είναι δύσκολο να αμφισβητήσουμε το σύστημα με τον τρόπο αυτό που προτείνει. Μπορούμε δηλαδή να, να καθορίσουμε τον ρόλο των ανθρώπων μέσα στις περιφέρειες, για παράδειγμα το άρθρο 84, έχουμε το κριτήριο για την διάκριση των περιφερειών. Αν έχω για παράδειγμα μια μεταβατική περιφέρεια με υψηλότερη ανεργία, θα πάρει περισσότερα χρήματα από μια περιφέρεια με λιγότερη ανεργία. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο άρθρο 84. Και ίσως εκεί μπορούν να συμπληρωθούν και άλλα πράγματα για να μπουν κάποια κριτήρια της επιλεξιμότητας. Με ενισχυθεί δηλαδή το κριτήριο της επιλεξιμότητας, αλλά δεν μπορεί να μπει σε αυτό, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να φύγουν από τη μέση περιφέρειες και να πει αυτά ισχύουν για όλους. Επίσης δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη διαγραφή του κώδικα διοντολογίας. Δεν βλέπω άλλωστε και το νόημα. Αφενός είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται διακρίσεις να εκπροσωπούνται και να μπορούν να επηρεάσουν τον σχεδιασμό. Αν όμως διαγραφούν, αν όμως ε, περικοπούν όλα τα κονδύλια τα οποία τους επιτρέπουν αυτή την ε, πρόσβαση, τότε ε, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό. Είναι επίσης κατά του αποθεματικού απόδοσης. Λέει ότι αυτό σημαίνει παραπάνω γραφειοκρατία. Εγώ όμως νομίζω ότι πρέπει να επιβραβευθούν οι περιφέρειες οι οποίες στείνουν στα πόδια τους καλά προγράμματα. Συμφωνώ βέβαια ότι η αναστολή των πληρωμών ασφαλώς αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος στην επιβράβευση αλλά όχι στην τιμώρηση ας πούμε έτσι. Και ξεκινάει και επίσης και από μια αιρεσιμότητα εκ των προτέρων, μια εξάντε conditionality. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πρώτα ένα πρόγραμμα. Πώς θα λάβει ο άνθρωπος με αναπηρίες τη δυνατότητα να μπορέσει να ενταχθεί αυτόνομα στην ε, εργασία, στην αγορά εργασίας. Χωρίς τα χρήματα δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό. Αυτό λέει η εξάντη conditionality. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να συμφωνήσω με τις τροπολογίες του κ. Κόσα. Σας ευχαριστώ κύριε Κέντς στα Ουγγρικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω στα Ουγγρικά για να μιλήσω στην κοινή γλώσσα που έχουμε με τον Άνταμ και να αξιοποιήσω όλα τα πλεονεκτήματα που μου προσφέρει η μετρική μου γλώσσα. Πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή ε, του Άνταμ Κοζά εμφανίζονται πολύ σημαντικά ζητήματα το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης εναρμονίζεται με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα χρειαστεί λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ στενά ώστε να εμφανίζονται οι ίδιες πτυχές και στα δύο κείμενα. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε επικοδομητικό διάλογο. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις, όπως έκανε και για το κοινωνικό ταμείο. Και σε αυτή την έκθεση βλέπουμε τη σύγκριση, τον παραλληλισμό με τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα άλλα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, ε, ένταξης των Ρωμά, απασχόλησης, ε, όχι μόνο με τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα, ώστε αυτό το ταμείο να χρησιμοποιηθεί, αυτά τα ταμεία να χρησιμοποιηθούν με τρόπο εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και εγώ διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά ότι υπάρχουν τροπολογίες ε, οι οποίες αφορούν τους ε, αναπήρους θα χρειαστεί να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των ατόμων και των ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Επίσης ε, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο κείμενο ενδεχομένω ε, το γεγονός ότι αυτά τα ταμεία δεν θα πρέπει να ενισχύουν τις ανισότητες ε, καθιονδήποτε τρόπο. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα ταμεία ε, δεν συνέβαλαν στην εξάλληψη της ε, ένδυας, στην εξάλληψη των περιπτώσεων εγκατάλειψης του σχολείου. Επίσης θα ήθελα να αναφέρεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η συμπληρωματικότητα διότι έχουμε διαπιστώσει ότι συχνά η χρήση των ταμείων είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει αυτή η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφορών ταμείων. δεν θα πρέπει να είναι αδύνατη αυτή η επικάλυψη. Συνεπώ αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε με τον Αντάμ Κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Αντάμ Κωσάκη για την εργασία του. Λέει κυρία Μωράν Σαρτιέ, οι τροπολογίε του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε όπως είπαν και οι συναδελφοί μου. Δεν θα επανέλθω σε αυτό, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για τη μέθοδο εργασίας μας. Βλέπουμε καλά ότι και οι δύο εκθέσεις είναι εξαιρετικά αλληλοσυμπληρωματικές και θα πρέπει να συντονιστούν η μία με την άλλη, ώστε οι συστάσεις οι συστάσεις της μίας υπάρχουν και στην άλλη, να μην υπάρχουν κενά μεταξύ τους και όλα αυτά να εμφανίζουν απόλυτη συνοχή. Προτείνω λοιπόν η ομάδα εργασίας του κυρίου Κόσα, οι συγητής και σκιώδεις συγητές και η ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που έχει ήδη συσταθεί να συνεργαστούν κάποια στιγμή για μια κοινή ανάγνωση και για τις δύο εκθέσεις, ώστε να είμαστε απολύτως βέβαιοι τι θα δείξουμε εμείς ως ε, Επιτροπή Απασχόλησης, διότι εν τέλει το θέμα δεν είναι, κάτι, δεν είναι θέμα πολιτικών ομάδων. Βλέπουμε ότι όλοι μαζί ε, βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Είναι η δική μας εργασία σε σχέση με το αποτέλεσμα της εργασίας των υπολείπων επιτροπών. Όπως έλεγε η κυρία Μπερές ε, προηγουμένως πριν ε, φύγει από την αίθουσα, πιστεύω ότι όλοι θα κερδίσουμε αν αφιερώσουμε λίγο χρόνο για κοινή εργασία. Σε κάθε περίπτωση αυτό προτείνω εγώ ως μέθοδο εργασίας. Äh, Εσείς κύριε Κώσσα θέλετε να λάβετε το λόγο στο τέλος ε, της συζητήσεως αυτής. Καλά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για τις παρεμβάσεις σας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που άκουσα από εσά συγκεκριμένες προτάσεις. Με γνωρίζετε ήδη. Έχετε ήδη δει στην βάση της εργασίας που έχω ήδη επιτελέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι λαμβάνω υπόψη τις απόψεις των διαφόρων συναδέλφων μου στα σχέδια γράφων που συντάσσω. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις. Γιατί προτείνω την κατάργηση του κώδικα συμπεριφοράς ή ιδεοντολογίας. Μου τέθηκε μια σχετική ερώτηση. Δεν με απασχολεί τόσο ο κώδικας. Σύμφωνα με το σχέδιο, διότι η εφαρμογή των προγραμμάτων ακόμη σε εκείνο το στάδιο δεν είναι ξεκάθαρη για τις χώρες μέλη. Δεύτερο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει το σχέδιό μου ότι οι ομάδες εργασίας συνεργάζονται. Ε, βλέπω ότι υπάρχει μια διαφορά απόσταση ανάμεσα στις προθεσμίες για την κατάσταση τροπολογιών, ενώ δεν υπάρχει δυσκολία να συνέλθουν οι δύο ομάδες για να εξετάσουν ενδεχόμενες προσαρμογές των τροπολογιών για να λάβει πιο ξεκάθαρη μορφή η εργασία αυτή. Νομίζω ότι τα δύο κείμενα πρέπει να απηχούν την ίδια θέση και αυτό είναι σημαντικό για την έκθεση. Αναμένω λοιπόν τις τροπολογίες σας, τις προτάσεις σας Ευχαρίστως να κάνετε προτάσεις. Εγώ ίδιος εργάστηκα με τρόπο θαραλέο, μπορώ να το πω ίδιος. Και γνωρίζετε ότι ίσως έχω τονίσει περισσότερο το πρόβλημα των προσώπων με αναπηρίες. Νομίζω όμως ότι είναι ευκαιρία να το θέσουμε εδώ και νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες και των άλλων ε, προσώπων που ε, αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Η Προεδρεύουσα, κυρία Χίρς, ευχαριστώ για τις τελευταίες σας παρατηρήσεις. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή. Την, αρμόδια, την αρμοδιότητα μάλλον εξουσίας έχει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εμείς ως απασχόλησης ζητήσαμε τη συμμετοχή μας σύμφωνα με το άρθρο 5051 αλλά δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Στις 23 Μαρτίου λέει πρόεδρος, 23 Μαΐου ενώ, 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι λίγη προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών και στις 10 Ιουλίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχολήσεως. Για απόψη σας ευχαριστώ.